Uh, Κυρίε και κύριοι, σχεδόν όλε οι πολιτικέ ομάδε εκπροσωπούνται. Οπότε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μα. Πριν περάσουμε στον δέκατο σημείο, τη συζήτηση με τον ε, Υπουργό Διομηχανία τον Μιγγέλ Σεμπαστιάν Πασκόν, να σας πληροφορήσω ότι ως συνήθως ε, στις συνεδρίες των συντονιστών που έλαβε χώρα το πρωί <clears throat> μετά την τακτική μας συνεδρίαση καταγράψαμε τα πρακτικά τα οποία θα μοιραστούν και ως το τέλος της σημερινής συνεδρίασης το απόγευμα εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Στα αριστερά μου έχω τον σημερινό μα προσκεκλημένο, τον Υπουργό της Ισπανική Κυβέρνησης για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και το εμπόριο, τον κύριο Μιγγέλ Σεμπαστιάν, ο οποίος εκπροσωπεί την, πρόοδη, την ασκούσα προεδρία του Συμβουλίου. Θα τον ακούσουμε σε σχέση με τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στα θέματα εμπορικής πολιτικής. Σας καλωσορίζω κύριε Σεβαστιάν Γκασκόν στην αρχή αυτής της Ισπανικής Προεδρίας όπου θα πρέπει εσείς να αναλάβετε την ευθύνη των πρώτων μιλών υλοποίησης της συνθήκης της Λισαβόνας. Η Ισπανική κυβέρνηση θα εγκαινιάσει τις νέες συνταγματικές διευθετήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Κατά τα άλλα, η συνθήκη της που επέφερε κάποιες αλλαγές επίσης αύξησε τις εξουσίες του Κοινοβουλίου. Θα περάσουμε λοιπόν στην αυτή διαδικασία με μεγάλο ενδιαφέρον για να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και εγώ ίδιο θα λάβω μέρος σε γεύμα της Επιτροπής Εμπορικής Πολιτικής. Νέο όνομα της πρώην Επιτροπής του άρθρου 133. Αυτά στι 12 Φεβρουαρίου φέτο. Για μας θα είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε την ομιλία σας, να ακούσουμε τις προτεραιότητες της Ισπανικής Κυβέρνησης και Προεδρίας για το πώς βλέπει το Συμβούλιο αυτή τη νέα φάση. Ενώ υπάρχουν και ζητήματα που πιέζουν, όπως ο γύρος διαπραγματεύσεων της ΔΟΧΑ στον ΠΟΕ. Οι διμερείς διαπραγματεύσεις για τις ε, συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών και η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ε, Νότιο Κορέα, την Λατινική Αμερική την Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα, τον Καναδά, τις Πολιτείες και το καθεξής. Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι η παρουσίασή σας θα μας οδηγήσει σε ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. με τα μέλη που θα θίξουν τα ζητήματα αυτά που θα βρίσκονται στους επόμενους 6 μήνες στην καρδιά τη επικαιρότητα για την Ισπανική Προεδρία. Σα καλωσορίζω και σα δίνω το λόγο. Uh, έχετε 10 λεπτά για την ομιλία σα και αμέσω μετά θα έχουμε συζήτηση και θα έχετε ξανά την ευκαιρία να απαντήσετε στα σχόλια των συναδέλφων. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, μέλη τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έχω την τιμή να μου δίδεται η ευκαιρία να εμφανιστώ μπροστά σας και να σας εξηγήσω το περιεχόμενο του προγράμματος που έχει προετοιμάσει η κυβέρνησή μας σε θέματα διεθνούς εμπορίου για την ε, Ισπανική Προεδρία. Πρόκειται για ένα εξάμεινο το οποίο θα είναι το εξάμεινο των μεγάλων αλλαγών σε θεσμικά θέματα όπως είπε και ο Πρόεδρος, μετά τέσσερις ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας. Μία νέα θεσμική αρχιτεκτονική στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσείς δηλαδή, που είστε το μοναδικό θεσμικό όργανο που εκλέγουν άμεσα οι πολίτες, ειδική βαρύτητα στα πλαίσια της δημοκρατικής νομιμότητας των αποφάσεων που εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια του Εθνούς Εμπορίου, η συνήθις ε, νομοθετική διαδικασία θα είναι η συναπόφαση. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η σύναψη διεθνών συμφωνιών θα απαιτεί και τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα πρέπει έγκαιρα να γνωρίζει ποια είναι η όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Η κυβέρνηση μου, λοιπόν, βλέπει πάρα πολύ θετικά το γεγονός ότι στα πλαίσια της ε, νέας συνθήκης Λισαβόνας θα υπάρχουν ε, ε, εξουσίες του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας στα πλαίσια τους ε, συνθήκης της Λισαβόνας και με τις δύο επόμενες προεδρίες έχει εκπονήσει το πρόγραμμα εργασίας του τους επόμενους 18 μήνες κυρίως προσπαθώντας να ευνοήσει το άνοιγμα των εμπορικών συναλλαγών. Οι τρεις προεδρίες έχουν καταρτήσει ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε δύο διπλές προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα, πρόθεσμα να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες, ώστε οι ευρωπαϊκές οικονομίες να ξεπεράσουν το συντομότερο δυνατόν την παρούσα κατάσταση οικονομικής στασιμότητας και να μειώσουν τις επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο. Απ' την άλλη, και πιο μακροπρόθεσμα, να θέσουμε τις βάσεις για να δώσουμε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία τις δυνατότητες μιας πιο ε, ισοσκελισμένης αηφόρου ανάπτυξης και πιο επωφελού για όλους. Και διάρκεια αυτού του εξαμήνου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το διεθνέ εμπόριο ένα από τα βασικά στοιχεία της ευημερία δημιουργής νέων ε, θέσεων απασχόλησης και της οικονομίας στις κοινωνίες μας που το απαιτούν. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε όλοι το σύνθημά μας που είναι περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες με λιγότερους φραγμούς. Αυτό το εξάμεινο θα καταβάλουμε σημαντική προσπάθεια σε πολυμερές επίπεδο. Γι' αυτό και ακολουθώντας τις τελευταίες ανακοινώσεις των ηγετών του G20 θα εργαστούμε ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του γύρου της ΔΟΧΑ με μια σφαιρική, φιλόδοξη και ισοσκελισμένη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι διατηθειμένοι να συμμετάσχουν με υποοικοδομητικό τρόπο στην επόμενη συνάντηση του ΠΟΕ που προβλέπεται για τα τέλος του μηνός Μαΐου. Το στόχος μας είναι παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την συμφωνία ε, εφέτος για να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο γύρος αυτός συνομιλιών της Δόχας εφέτος. Επίσης πρέπει να πω ότι θα ενισχύσουμε και τις διάφορες και θα προωθήσουμε τις διάφορες διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση νέων κρατών στον ΠΟΕ, όπως Φερρυπίνη, η Ρωσία, η Λιβύη, η Βοσνία, Ζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Έτσι θα ενισχύσουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα και θα θέσουμε τις βάσεις ε, με καλύτερο τρόπο για να βελτιώσουμε και τις διάφορες διμερείς εμπορικές ε, σχέσεις μέσω συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου. Εξάλλου, όσον αφορά την ε, περιφερειακή ε, διάσταση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πω ότι θα συνεχίσουμε και εδώ τις διάφορες διαπραγματεύσεις. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Λατινικής Αμερικής, θα εργαστούμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αρκετά σύντομα τις διάφορες διαπραγματεύσεις που έχουμε με την ε, κοινότητα των άνδρων Κεντρική Αμερική. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις πριν από την σύγκληση της διάσκεψης ε, κορυφής ε, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής με την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο. Η πρόθεσή μας είναι όταν θα μπορέσει να ξεπεραστεί η κρίση στην Ονδούρα, να ολοκληρώσουμε την συμφωνία σύνδεσης με τους χώρες της Κεντρικής Αμερικής για να ε, βοηθήσουμε περισσότερο την ε, εμπορική ενσωμάτωση στην ε, κοινή Αμερικής. Συμπληρωματικά είναι προτεραιότητά μας να ολοκληρώσουμε τις συμφωνίες διαπραγμάτευσης με την Κολομβία, το Περού και ίσως και με το Εκουαδόρ καθώς που είναι ε, μέλη της ε, κοινότητας των Άνδεων και να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε τις διαπραγματεύσεις το, σε συμφωνία σύνδεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μερκοσούρ. Και σε σχέση με το Μερκοσούρ πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την συμφωνία που αφορά 700 εκατομμύρια άτομα στην περιοχή εκείνη. Θα ε, ενισχύσουμε την οικονομική ε, ενσωμάτωση, θα προωθήσουμε το εμπόριο και τις ε, επενδύσεις επίσης στην ευρωμεσογειακή περιοχή. Δημερός, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω την ε, πρόσφατη ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων συμφωνίας ελεύθερου πορείου με την Κορέα. Πρόκειται για πολύ σημαντική συμφωνία και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει τον Φεβρουάριο η Επιτροπή να παρουσιάσει προς υπογραφή μια πρόταση στο Συμβούλιο στην Ασία η Ινδία και η Κίνα αναμφίβολα είναι δύο πάρα πολύ ενδιαφέρουσε αγορές για το Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια του 2010 θέλουμε να προχωρήσουμε ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία και στην ανείχνευση νέων οδών επανισορρόπηση τη διμερούς σχέση μα με την Κίνα. Όσον αφορά τη Ρωσία, ο κύριο στόχο μα είναι να διευκολύνουμε την προσχώρησή τη στην ΠΟΕ. Μιλούμε για ένα στρατηγική σημασία εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερο για θέματα ενεργειακά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχη συγκεκριμένη περίπτωση η διαπραγμάτευση ενός νέου συμφώνου πλαισίου. Επίσης πρέπει να πω ότι τα ενεργειακά θέματα είναι μέρος σημαντικό της συμφωνίας η οποία διαπραγμα... την οποία διαπραγματευόμαστε με την Ουκρανία. Η δημιουργία μιας ζώνης ελευθέρου εμπορίου θα συνεισφέρει στην ε, προοδευτική ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενισχύσει τη νέα στρατηγική της ε, ανατολικής σύνδεσης. Εξάλλου, ένας από τους στόχους προτεραιότητες μας είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις οικονομικές μας σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό θα ενισχύσουμε το ΤΕΚ που είναι ένα μέσο χρήσιμο και αποτελεσματικό για την ανείχνευση και την ε, κατάργηση των ε, μη τελωνιακών φραγμών που δυσκολεύουν τις ε, εμπορικές ροές και τις διμερείς επενδύσεις. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο, η, επίσης σημαντικό είναι, η, σημαντική είναι η οικονομική και εμπορική συμφωνία που πρέπει να συνάψουμε τον Καναδά. Θα θέλαμε, εκτός από τα διάφορα θέματα τα οποία θα εξετάσουμε διμερός, πολυμερός και περιφερειακά, να πούμε ότι θα πρέπει μέσω πρόθεσμα να ξαναθέσουμε τις βάσεις μία κοινή εμπορικής πολιτικής. Γι' αυτό θέλουμε να υπάρξουν συζητήσεις και υποδείξεις και σχόλια για τις στρατηγικές γραμμές που θα πρέπει να ε, ε, είναι οι γενικές γραμμές πλεύσεως της πολιτικής μας τα επόμενα πέντε χρόνια. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τη στρατηγική πρόσβαση στις αγορές, ώστε να μην υπάρχουν πειρασμοί προστατευτικοί. Στα πλαίσια όλων αυτών των ε, πολιτικών που θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε, ε, προτείναμε στην Επιτροπή να καταρτήσει ένα εγχειρίδιο δράσης για να συστηματοποιούνται οι δράσεις που πρέπει να, να πραγματοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίση θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο άνοιγμα των αγορών δημοσίων ε, και κρατικών προμηθειών και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Μία άλλη από τις ε, προτεραιότητές μας είναι να μπορέσει να συναυθεί η εμπορική συμφωνία κατά της παραποίησης, η λεγόμενη ACTA. Πρόκειται για μία συμφωνία η οποία θα αποτελέσει και διάρκεια τη δική μα Προεδρία το αντικείμενο δύο γύρων διαπραγματεύσεων. Εξάλλου, η κυβέρνησή μα θεωρεί ότι το εμπόριο είναι ένα βασικό μέσον για την πρόθεση τη ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τους ε, ποιοτικούς στόχους στόχους χορήγησης βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, η βοήθεια που παρέχεται στον τομέα του εμπορίου από, το από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέρχεται σε 2 δις ευρώ ετησίως. η Ισπανική Προεδρία να λαμβάνει τη δέσμευση να συνεχίσει να συνεργάζεται με την Κομισιό και τα κράτη-μέλη, ώστε αυτή η βοήθεια να συνεχίσει να είναι βοήθεια ποιοτική, ώστε να υλοποιήσουμε τον τελικό μας στόχο, που είναι η διευκόλυνση των ε, αναπτυσσομένων χωρών, ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει η συμμετοχή τους στο πολυμερές σύστημα εμπορίου. Επίσης, θα ήθελα, τελειώνοντας, να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για να μπορέσει να συναυθεί η Διεθνή Συμφωνία για το Εμπόριο Όπλων στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και τη συμμετοχή μας στις διαπραγματεύσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του ΩΣΑ. Τελικά, θα πρέπει να σας πω ότι προβλέπουμε ε, και κάποια δράση τους επόμενους ε, μήνες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τις κλιματικές αλλαγές, την ε, όλο και αυξανόμενη σχέση μεταξύ εμπορικής πολιτικής και ενεργειακής πολιτικής, υγείας, κοινωνικών ε, δικαιωμάτων, προστασίας του καταναλωτού και ισότητας μεταξύ των δύο. Τελειώνοντας κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου αντιμετωπίζει το εξάμεινο της Προεδρίας με μια ευρύτατη ατζέντα στην οποία υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση υπεύθυνη, σταθμισμένη, σε, έχοντας επιτύχει συμφωνίες μεταξύ μας, ώστε να μπορέσει το διεθνές εμπόριο να εκδίδει ένας από τους κύριους φορείς ανάπτυξης και αηφορίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γι' αυτό θα εργαστούμε και υπολογίζουμε και στην δική σας βοήθεια όπως και σε άλλα θέματα μετά από την ε, θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε για αυτή τη σαφή παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Πρώτον, ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Ο κύριος Σάλπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη τιμή σας καλωσορίσουμε εδώ. Ως Ισπανής θα ήθελα να σας ευχηθώ επιτυχία. Επιτυχία σας θα είναι και της Ισπανίας και της Ευρώπης επιτυχίας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στην ε, ε, συμφωνία την οποία έχει διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Νότια Κορέα. Εμείς θα θέλαμε να εμβαθυνθούν οι σχέσεις μας με αυτή, την σχέση, με αυτή τη χώρα της Ασίας. Και αυτό νομίζουμε ότι θα είναι επωφελέ και για τι επιχειρήσει τη Νοτιού Κορέα και για τι δικέ μα. Πρέπει να σα πω ότι εμεί στο ΕΛΚ υποστηρίζουμε. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ το ελεύθερο εμπόριο. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην δημιουργηθούν μειονεκτήματα για κάποιες ε, βιομηχανίες της Ευρώπης, κυρίως για την αυτοβιομηχανία διότι ξέρετε ότι πάρα πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι εξαρτώνται από την αυτοκίνητο βιομηχανία. Ξέρουμε ότι κυρίως στη δική μας τη χώρα βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό τα αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάζονται στην Ισπανία με αυτά που κατασκευάζονται στην Νότια Κορέα. Ξέρετε πόσο υψηλό είναι το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας. Ε, θα ήθελα να μου πείτε αν συμμερίζεστε κι εσείς αυτές τις ε, ανησυχίες τις οποίες εκφράζω και ποια είναι τα βήματα τα οποία θα κάνετε για να μπορέσετε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα και να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω, ε, σας ε, απασχολεί το τι θα γίνει μόλις συναυθεί αυτή η συμφωνία με την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ισπανία. Επίσης, αναφέρατε την συμφωνία ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής ε, Αμερικής. Είπατε ότι ενδεχομένως θα συναυθεί αυτή η συμφωνία στις 18 Μαΐου στο Μάιο. Αυτό σημαίνει ότι εσείς αυτή τη στιγμή αναγνωρίζετε την κυβέρνηση της Τεθιού Γάλπα. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των ε, σοσιαλιστών, ο κύριος Μενέντες. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή μας. Είπατε και τονίσατε πόσο σημαντικό είναι για την Προεδρία η σύναψη συμφωνιών με τη Μερκοσούρ, με την κοινότητα των Άνδρων και με την χώρε Κεντρική Αμερική. Θα ήθελα συγκεκριμένα να σα ρωτήσω το εξή για το Μερκοσούρ. Σήμερα το πρωί μα επισκέφθηκε ο πρέσβη τη Βραζιλία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά από πέντε χρόνια Ε, στασιμότητα των διαπραγματεύσεων δεν φαίνεται να είναι τα πράγματα πάρα πολύ ε, σαφή. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες ε, σοβαρές δυσκολίες που ίσως μας εμποδίσουν να καταλήξουμε συμφωνία. Επίσης, όταν αναφέρει συμφωνίες σύνδεσης, όχι με την Κεντρική Αμερική, ο κύριος Θάλμπα ανέφερε το θέμα αυτό και σας μίλησε για κάποιες δυσκολίες, συγκεκριμένα την κοινότητα των Άνδεων. Πιστεύετε ότι εκ μέρους των πιο αντιδραστικών κρατών ε, της Βολιβίας και του Εκουαδόρ ε, στις διαπραγματεύσεις αυτές φαντάζεστε ότι θα δημιουργηθούν περισσότερα προσκόμματα από τον ένα σε σχέση με τον άλλο. Ευχαριστώ εκ μέρους του Άλντε. Ο κύριος Καζάκ ζητά το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε όταν ε, η αντιπροσωπεία μας ε, είχε επισκεφθεί την Ισπανία και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω ε, εδώ με την αρχή της Προεδρίας. Θα ήθελα σαν επικεφαλής της Προεδρίας ε, που ασχολείται με τα θέματα μας να αναφερθώ εις την ρύθμιση της αγοράς σημαντικών προϊόντων διότι στο παρελθόν η Ισπανία ήταν υπέρ μίας τέτοιας πρότασης το 2009 είχαμε ε, ε, ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αυτό το πνεύμα και στη συνέχεια υπήρξαν ε, τρεις εναλλακτικέ προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις οποίες συζητήσαμε ε, αλλά Έκτοτε ε, επανήλθαμε στην αρχική πρόταση. Ε, μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι ε, θα ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία επί της Προεδρίας σας και τι θα χρησιμοποιήσετε σαν μέσον για να επιτύχετε συνένεση. Δεύτερον, όταν είχαμε επισκεφτεί την Ισπανία τον Νοέμβριο μας είχατε πει ότι δεν πρόκειτο να ασχοληθείτε, ότι ε, θεωρούσατε ότι έχει λυθεί ε, το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τι γίνεται όμως με τις συνδικαλιστικές ε, οργανώσεις. Η θέση της Προεδρίας σας παραμένει η ίδια είναι όλες οι κυβερνήσεις ομόφωνες ότι υπάρχει μία θετική αντιμετώπιση ή μπορεί να υπάρξει μία μειονότηση η οποία θα μπλοκάρει το θέμα και τι θα γίνει με τις εφαρμοστικές διατάξεις. Υπάρχει περίπτωση ένας τέτοιος κανονισμός να υιοθετηθεί προτού ε, εγκριθεί η συμφωνία από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την ε, παρέμβασή σας ε, και σας χαιρετίζουμε για την πρωτοβουλία σας να συσφίξατε τις σχέσεις με την Λατινική Αμερική και το συμπέρασμα της παρεμβάσεώς σας ότι χρειάζονται ε, πρωτοβουλίες για να συνδυάσει κανείς τα κοινωνικά δικαιώματα με το περιβάλλον, με την διατροφική ασφάλεια και τα υπόλοιπα θέματα που εκκρεμούν. Θέλω να ρωτήσω το εξή Στο θέμα του κλίματος, θα μπορούσε η Ισπανία να προτείνει μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μεταφορά τεχνολογίας για να διευκολύνει αυτές τις μεταφορές κατά τρόπο ώστε οι νότιες χώρες να έχουν πιο καθαρές παραγωγές. Επίσης η Προεδρία της Ισπανίας έχει προσυπογράψει ε, την έκθεση του ε, γραμματέα ε, Τζον Ρούγκη εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα μέτρα τα οποία σκοπεύετε να πάρετε διότι θέλατε μία συμφωνία. Μία συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις Ονδούρες. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε ότι η θέση της Ισπανίας στη Σύνοδο ε, με τη Λατινική Αμερική το Νοέμβριο αλλάζει. Αναγνωρίζετε το κυβέρνηση που προέκυψε από πραξικόπημα. Και επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζετε ότι εδώ συζητούμε συχνά την κατάσταση της Κολομβίας που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως ως τώρα η Ευρώπη. Δυστυχώς κατά την άποψή μας δεν έλαβε επαρκείς πρωτοβουλίες για να προβλέψει το πολιτικό το αυτό ζήτημα του σεβασμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας δώσετε τη γνώμη σας επ' αυτού και όσον αφορά την Ευρωμέντ η αξιολόγηση των επιπτώσεων για την ε, ε, επιβεβαίωση αυτής της συμφωνίας ήταν πολύ αρνητική όπως και οι μελέτε των επιπτώσεων για συμφωνίες με τη Λατινική Αμερική. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε σχετικά με αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και πόσο θα τα εντάξετε στο γενικότερο πλαίσιο της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλώ εν ονόματι του κυρίου Στέρντι αλλά θα μιλήσω τσέχικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίασή σας διότι ε, θίξατε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και είπατε ότι πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και στηρίζω αυτή την άποψη, ε, συμφωνώ απολύτως. Ε, εκπλήσωμαι και θαυμάζω το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμά σας σχετικά με τη συμφωνία με το Μερκοσούρ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία ε, στην ολοκλήρωση των συμφωνιών, διότι νομίζω ότι ο τομέας αυτός είναι πάρα πολύ πολύ Θέλω όμως να σας κάνω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, ε, ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα. Σαν Προεδρία Πώς θα αξιολογήσετε την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με ε, την Σρι Λάνκα και επιπλέον υπάρχει πίεση να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέτρα και σε άλλες χώρες. Πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρούμε αιτιολογημένη αυτή την, ε, ε, ε, την πρόθεση. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο ίσως συνδυάζεται με το γεγονός ότι στην Ισπανία υπάρχουν μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ εδώ εκπροσωπείται το Συμβούλιο. Για πέστε μας πώς αξιολογείται την ε, συμφωνία για ε, την συνεργασία μεταξύ, ε, ελεύθερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Κορέας. Θέλετε να παρέμβετε τώρα? Ωραία. Ο κύριος Σόλτς. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θέλω να προσθέσω ορισμένα ερωτήματα σε αυτά των συναδέλφων, ιδίως όσον αφορά τις ε, συναλλαγές με το Μερκοσούρ. Ε, δηλαδή συγκεκριμένα ε, περαιτέρω και με τη συμφωνία με την Κολομβία, με την Ονδούρα. Πώς εσείς αξιολογείτε τις δυνατότητες δεδομένων των συγκεκριμένων προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προβλημάτων των ανθρώπων να μπορέσουν να έχουν μία ε, ε, καλή διαβίωση, να ε, διατηρηθούν αυτά τα δικαιώματα. Επιπλέον, όσον αφορά τις συζητήσεις με τον Καναδά που έχουν ξεκινήσει και ε, ε, αποβλέπουν να τελεσφορήσουν ε, ο Σονούπο έχετε συγκεκριμένες φιλοδοξίες και πλέον πώς βλέπετε τις σχέσεις με την Κούβα. Αυτές είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Υπάρχουν και άλλοι που ζητούν το λόγο, αλλά θα αφήσω για ένα δεύτερο γύρο και δίνω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ισπανίας για να απαντήσει στις ερωτήσεις των πολιτικών ομάδων. Για ένα δεκάλεπτο, γιατί μετά θα υπάρξει και δεύτερος γύρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζοντας θα αναφερθώ στην συμφωνία με την Κορέα που ανέφερε τόσο ο κύριος Θάλμπα όσο και ο κύριος Σάκαλ. Από τη δική μας άποψη η συμφωνία με την Κορέα είναι καλή συμφωνία. Πιστεύουμε ότι περιέχει ρήτρε προστασίας από καταστάσεις ανισορροπίες διότι οι μεταβατικές περίοδοι μεταξύ άλλων μας επιτρέψει να προστατευτούμε από την φιλελευθεροποίηση μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στον τομέα και να ξεπεραστεί η κρίση. Και υπάρχουν δυνατότητες ε, εμπορικών συναλλαγών με πάρα πολλές επιχειρήσεις, πάρα πολλών τομέων από την Ευρώπη, στον τομέα της βιομηχανίας, στον τομέα των υπηρεσιών, ίσης όρης, για να μην πω καλύτερα, πότε βρίσκονται αυτή τη στιγμή σχέση με την Κορέα οι ανταγωνιστές μας ή είπα όσον αφορά τις κρατικές προμήθειες πρέπει να πω ότι έχει η θέση μας βελτιωθεί πολύ σημαντικά. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράσουμε ότι αν ε, σε κάποιους τομείς αυξηθεί στην εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά ο ανταγωνισμός η... το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καθαρή βελτίωση διότι θα υπάρχουν περαιτέρω επενδύσεις, εμπορικέ συναλλαγέ και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τώρα, στα πλαίσια αυτή τη συμφωνία θα ήθελα να αναφερθώ όλου ιδιαίτερω στον τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία. Έγιναν σχετικά δύο σχόλια. Πρέπει να πω ότι η διαπραγμάτευση αυτής ε, της συμφωνίας έλαβε υπόψη τα συμφέροντα τη ευρωπαϊκής Αυτοκινητοβιομηχανία, δεδομένου ότι προβλέπονται κατάλληλε περίοδοι ε, προσαρμογής όσον αφορά την ε, κατάργηση μη τελωνιακών φραγμών ώστε να μην πληγεί η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Όπως σας είπα θα υποστηρίξουμε και θα εγκρίνουμε την ε, σύναψη αυτής της συμφωνίας βεβαίως σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιό σε πλαίσιο διαφάνειας και συμμετοχής όλων έτσι όπως προβλέπεται από την συνθήκη της Λισαβόνας. Σε σχέση με την ε, Κεντρική Αμερική και την ερώτηση την πολύ συγκεκριμένη για την Ονδούρα θα πω ότι η Ισπανική κυβέρνηση πιστεύει ότι μετά από τη λήψη των καθηκόντων του νέου Προέδρου θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις της χώρας αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορέσουμε να θέσουμε και πάλι σε εκκίνηση την διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Σύνδεση με την Κεντρική Αμερική, η οποία ελπίζουμε θα μπορέσουμε να ρεκριθεί του επόμενου μήνε. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μια δύσκολη κατάσταση, αλλά προσπαθούμε με κάθε τρόπο να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας. Όσον αφορά τώρα την ε, κοινότητα των Άνδεων, έγιναν πολλά σχόλια και ερωτήσεις. Ένα από αυτά αφορούσε όλος ιδιαίτερος τον αποκλεισμό ή όχι των κρατών των Άνδεων, που, της περιοχής των Άνδεων που δεν έχουν συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, κυρίως του Ισημερινού και της Βολιβίας. Πιστεύουμε ότι εμείς μια τέτοια πολυμερή συμφωνία δεν ε, αποκλεί κανέναν από τη διαπραγμάτευση. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι δεν συμμετείχαν στην διαπραγμάτευση, έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν σε συμφωνίες εμπορικού τύπου. Ιδιαίτερα όσον αφορά την Κολομβία, εμείς ε, πρέπει να πω ότι προσδίδουμε μεγάλη σημασία στην ε, εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και, μπορούμε, και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μπορέσουν να προσ να μπορούμε να προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εργαζομένων στην Κολομβία. Και πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να βρούμε αποτελεσματικούς θεσμικού τύπου μηχανισμούς που θα μας δώσουν την εγγύηση ότι δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση. Πρέπει να πω επίσης ότι και σε σύμπραξη με τον ΟΗΕ και με τον ΟΗΤΕ, σύμφωνα με, την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας, σύμφωνα με τις συμφωνίες οι οποίες έχουν ε, επιτευθεί. Υπάρχει σχετική εισήγηση ότι κάνει ό,τι μπορεί η Κολομβία για να προασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Υπήρξαν στο παρελθόν κάποια ε, προβλήματα, αλλά πρέπει να πω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και στις συμφωνίες που ε, έκανε με τη ΣΥΠΑ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι εμείς καλύτερα να έχουμε μία άποψη ε, συμπερίληψης παρά μία άποψη αποκλεισμού κάποιων. Αυτό το οποίο θέλουμε κυρίως είναι να διευκολύνουμε την πρόοδο ώστε να μπορέσουν τα ε, δικαιώματα όλων να γίνονται σεβαστά από όλους. Και πρέπει να πω ότι εμείς εάν θέλετε, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να επανέλθουμε για να μιλήσουμε για τα συνδικαλιστικά ε, δικαιώματα της Κολομβίας. Εξ ονόματος της κυβέρνησης λοιπόν και της Προεδρίας θα ήθελα να σας μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Μερκοσούρ. Το ανέφερε ο κύριος Μέντελ Δελβάλλη. Πιστεύουμε ότι θα προσπαθήσουμε στα πλαίσια της Προεδρίας, από τη μεριά μας ε, της Προεδρίας και από τη μεριά εκείνων της Αργεντινής, θα γίνει κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε διαπραγματεύσεις. Στην ε, διάσκεψη κορυφής του Εστορίλ το προηγούμενο Νοέμβριο, η πρόεδρος της Αργεντινής και οι υπόλοιποι οι ηγέτε, καθώς και ο δικός μας προηγούμενο είπαν ότι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις ώστε να μπορέσουν να ε, ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει για να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να εργαστούμε για να μπορέσει να συναφθεί αυτή η συμφωνία που όπως σας είπα για μας είναι η πιο φιλόδοξη και για τον κόσμο ολόκληρο δεδομένου ότι θα σημαίνει μεγάλη αύξηση των ε, ε, εμπορικών ροών και των επενδύσεων που θα αφορούν 700 εκατομμύρια άτομα. Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία με μεγάλη δυναμικότητα όσον αφορά μια εμπορική συμφωνία παγκόσμια. Και βεβαίως θα θέλαμε το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και τις διαπραγματεύσεις με το Μερκοσούρ. Αλλά αυτή τη στιγμή αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστέ, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα μπορέσει να συμβεί, τουλάχιστον κατά τη δική μα Προεδρία, αλλά θα θέλαμε να θέσουμε ένα πιο πραγματιστικό στόχο. Δηλαδή, να μπορέσουμε να επανενεργοποιήσουμε τι διαπραγματεύσει που, όπω ξέρετε κυρίε και κύριοι, βρίσκονται σε στασιμότητα, είναι μπλοκαρισμένες από το 2004. Θέλουμε λοιπόν να ξαναρχίσουμε αυτό τον διάλογο ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε, ένα, σε μια συμφωνία ισοσκελισμένη και σύμβατη με τους κανόνες του ΠΟΕ. Όσον αφορά το περιβάλλον και το εμπόριο, το περιβάλλον και το εμπόριο, είναι ένα ιδιαίτερα προσφυλές σε μας θέμα. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις υπάρχουσες για αυτό το τομέα πρωτοβουλίες. Θα αυξήσουμε τον αριθμό των κρατών που υποστηρίζουν τον κατάλογο των ε, προϊόντων που μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και η μετά την Κοπεχάγη και τον γύρο της Δόχα δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα τη διάρκεια της δική μας προεδρία, αλλά λογικά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε οποιαδήποτε τέτοιου είδους ε, τρέχουσα διαδικασία υπάρχει να την προωθήσουμε. Κύριε Καζάκ, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από την επίσκεψή σας στη Μαδρίτη που είχαμε πιο πολύ ζέστη από ό,τι σήμερα εδώ. Στο θέμα της ονομασίας προσέλευσης πιστεύω ότι βελτιώνονται οι πληροφορίες που δίδονται στον καταναλωτή με μεγαλύτερη διαφάνεια και έτσι, αλλά έτσι έχει ο καταναλωτής την επιλογή μεταξύ ενός πιο ακριβού πλην όμως ε, καλύτερου προϊόντος όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με ένα άλλο πιο φθηνό στο οποίο όμως δεν τηρούνται κάποιες ε, ε, αρχές. Θα πρέπει, δεν είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα, θα πρέπει να κάνουμε κάτι με πλήρη ε, σαφήνεια ώστε να μην δημιουργούμε σύγχυση στον καταναλωτή και κυρίως να μην δυσκολεύουμε την κατάσταση των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων. Θα πρέπει να αναθεωρήσει την πρότασή της η Επιτροπή για να μπορέσει να συγκεράσει όλα τα σημεία ε, τα οποία ενδιαφέρουν τα κράτη-μέλη και τα οποία ε, εμείς δείχνουμε ιδιαίτερη διευθυνσία. Συγγνώμη, άφησα κανένα θέμα απ' έξω. Ναι, την ε, Σρι Λάνκα. Ξέρουμε πόσα προβλήματα θα δημιουργήσει το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί με ε, την ε, Σρι Λάγκα. Ξέρουμε όμως ότι είναι πάρα πολύ σαφής ε, η κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να εφαρμόζεται με σαφήνεια, διαφορετικά το μέσο αυτό το οποίο διαθέτουμε θα χάσει οποιαδήποτε αξιοπιστία. Ε, το θέμα αυτό του συστήματος προτιμήσεων είναι ένα σύστημα το οποίο ε, προσφέρει πάρα πολλέ δυνατότητες στην κυβέρνηση της Σρι Λάνκα, αλλά πρέπει και εκείνη να συμμορφωθεί. Εάν λοιπόν ε, μπορέσει να ε, ακολουθήσει τους κανόνες, η Σρι Λάνκα θα συνεχίσει να επωφελείται από αυτό το μέσο. Τη στιγμή όμως ε, που η κυβέρνηση αναλάβει τις δεσμεύσεις και εφαρμόσει τις διάφορες ρήτρε αυτού του μέσου. Η Κούβα, και, εδώ με αυτό τελειώνω. Αναγγείλαμε τη διάρκεια της ε, Προεδρίας έχουμε την πρόθεση να κάνουμε μία εμπεριστατωμένη συζήτηση για να μπορέσουμε να σκιαγραφίσουμε τις γενικές γραμμές της πολιτικής μας με την Κούβα και να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να διαμορφώσουμε την ε, θέση της Ευρωπαϊκής ε, νοσής για αυτό το θέμα. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι κατά βάση πολιτικό και θα συζητηθεί και εκτός της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να σας ενημερώσω ότι έχει γίνει προσφορά από την Ισπανική κυβέρνηση να προσέλθει και ο αντιπρόεδρος της Ισπανικής κυβέρνησης. Η κυρία για την πρόταση τη Ισπανική κυβέρνηση. Κυρία Τερέζα Φερνάντε. Κυρία Ντελαβέγκα, η οποία θα μπορούσε να συζητήσει μαζί μας. Ας συνεχίσουμε όμως με το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Εδώ υπάρχει και το θέμα του χρόνου. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε 1,5 λεπτό, 2 λεπτά το πολύ ο καθένας. Βέβαια στο καταλόγο αγορητών, ο κύριος Μάρτιν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό για τις ειλικρινείς και ξεκάθαρες απαντήσεις του. Έχω ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα. Να πω ότι συμφωνώ μαζί σας για την Νότιο Κορέα οποιαδήποτε αξιολόγηση αυτής της Συμφωνίας ελευθερομπορίου πρέπει να γίνει βάση και των διεκδικήσεων τη Ευρωπαϊκής Ένωση και να συνεχίσουμε να τι επιδιώκουμε. Έπειτα για τι ΗΠΑ. Είπατε ότι είναι προτεραιότητα για την Ισπανική κυβέρνηση η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με τι ΗΠΑ. Εδώ χρειάζεται όμω διατλαντικό οικονομικό συμβούλιο για να το πετύχουμε κάτι τέτοιο. Και η συμμετοχή του. Το κείμενο έχει δείξει ότι είναι ελάχιστα επιτυχημένο τώρα. Θα συνεχίσουμε προ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν με το Διατλαντικό Συμβούλιο. Και αν ναι, σε ποια ακριβώ ε, προσέγγιση προσλέπετε. Έπειτα για την θέση στην Κολομβία ήσασταν πολύ ξεκάθαρο. Όμω, εδώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Η Κολομβία είναι μια από τι πιο επικίνδυνε χώρε ε, στον κόσμο δεν υποφέρουν μόνο οι συνδικαλιστέ στην ε, Κολομβία, αλλά και οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι γυναίκε που είναι θύματα του πολέμου, από επεισόδια και κρούσματα βιασμών και το καθεξής. Υπάρχει σοβαρό φαινόμενο βίας κατά των γυναικών εκεί. Έτσι λοιπόν, ε, πώ θα το δείτε αυτό το θέμα στα πλαίσια μια μιας συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Κολομβία. Λέτε ότι θα υπάρχει μια ρήτρα πολύ έντονη για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε μια τέτοια συμφωνία. Όμω, εγώ πιστεύω ότι να αποσπάσουμε τέτοια συμφωνία, το μόνο που θα γίνει είναι ότι η Επιτροπή θα κάνει μια πρόταση και το καθένα από τα κράτη-μέλη θα δεχτεί. 27 από του 27. Όσο έντονη και ρητή να είναι η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν αλλάζει τίποτα εφόσον υπογραφεί η συμφωνία. Είναι σχεδόν αδύνατο μετά τα πράγματα να αλλάξουν. Αυτό λοιπόν που σας ζητώ είναι να μην βιαστούμε. Να φέρουμε τους Κολομβιανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά πριν καταλήξουμε και υπογράψουμε τη Συμφωνία Ελευθερμπορίου, να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή τη χώρα περισσότερο. Ευχαριστούμε ο κύριος Κάσπαρη από το Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αφού έχουν συζητηθεί τόσα θέματα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αξιολογούν ότι η Κολομβία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με τη δεκαετία του 90. Αλλά έχω ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στη Νότιο Κορέα. Αλλά συγκεκριμένη ερώτηση. Μπορείτε να προχωρήσετε στο θέμα duty drawback με την Κορέα. Ε, θα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την πολιτική μας ομάδα. Επίσης ε, για τα εμπόδια για το εμπόριο διότι οι Κορεάτες δεν μειώνουν τους δασμούς. Μπορείτε να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θίξει το θέμα αυτό με τους Κορεάτες και πάλι. Επίσης, εάν κατάλαβα σωστά τη μετάφραση, είπατε προηγουμένως ότι προβλέπετε να κάνετε ε, ε, ένα νέο ορισμό της Μορικής πολιτικής μεσοπρόθεσμα και όταν κοιτάζω το πρόγραμμα της Προεδρίας σας βλέπω ότι και αναφέρομαι εδώ στο κείμενο το, ο ρόλος της εμπορικής πολιτικής σαν εργαλείου θα ενισχυθεί κατά την Ισπανική Προεδρία με εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ήξερα δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατυπώσει μία νέα, ε, μία νέα πολιτική στο εμπορικό τομέα. Δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο από τον κύριο Μπαρόζο θα θέλω λοιπόν να ξέρω τι μας περιμένει από εκεί. Και τρίτον, ε, ε, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Πιστεύετε ότι το Συμβούλιο θέλει ε, να βοηθήσει να μπορέσουν να συμμετάσχουν, να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Γιάννης από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας που μας επέτρεψε να διευκρινίσουμε πολλά θέματα. Πάρα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο θέσατε κάποια θέματα, αλλά θα ήθελα κάποιες περισσότερες εξηγήσεις για κάποια θέματα και να κάνω και πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις σε άλλα. Μιλήσατε για την δέσμευση να μπορέσουμε το 2 να ολοκληρώσουμε τον γύρο των συμιλιών της ΔΟΧΑ. Αυτή είναι η μητέρα των μαχών. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και συγκεκριμένο μου είναι είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά όχι επαρκής να υπάρχει συνοχή, συνένεση μεταξύ των 27, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Για να έχει σαφή εντολή στις ε, μελλοντικέ διαπραγματεύσεις του 2010 η Κομισιό. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, για το πώς υπάρχει πρόβλημα με τον ε, αυτοκινητόδρομο άρχα 400 μη στην Ανδαλουσία. Το κάνω αυτό όχι σε εσά ως Υπουργό, αλλά ως ε, βουλευτής της Σεβίλης. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Είπαν κάποιοι συναδελφοί σας ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει βία στην ε, ε, Κολομβία, ας μην την τιμωρήσουμε πάρα πολύ για να μην ε, χάσουν τη δυνατότητα να έχουν κάποια δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο και παρακαλώ δεχτείτε τις ευχές μου για καλή τύχη και επιτυχία στο εξάμενο της Προεδρίας. Τη ισπανική προεδρία. Ήθελα να παρέμβω, αλλά με φοβήσατε λίγο με τι απαντήσει σα, γιατί τουλάχιστον τρει συνάδελφοι έκαναν ερώτηση για την Νότιο Κορέα. Και εδώ υπάρχουν κάποιε αντιφάσει. Εσεί μιλήσατε με πολύ βεβαιότητα και... Ότι... και σιγουριά ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία πολύ σύντομα, πριν εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα πράγματα. Μας λέτε ότι 130 ευρωπαϊκά προϊόντα και βιομηχανίε εκπροσωπούνται στη χώρα, ενώ εμεί μαθαίνουμε ότι είναι τουλάχιστον 300. Επίση, μόλι είχαμε ένα νέο επίτροπο, τον κύριο Ντεκούχτ, ο οποίο είπε και χάρηκα ιδιαίτερα να τον ακούω, ότι τι ε, ρήτρε, τι σχετικέ ρήτρε θα τι δούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Λοιπόν και εσείς σκεφτείτε να μην βιαστείτε ότι μπορείτε να περιμένετε, να μελετήσετε καλύτερα το θέμα για να αποφύγετε τα επικριτικά σχόλια. Ευχαριστούμε και ο κύριο Λάγκη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, στο τέλος της πρώτης παρεμβάσεώς σας είπατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα το επίκεντρο της εμπορικής πολιτικής και αυτό με χαροποίησε ιδιαιτέρως. Εξού και η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής εσείς τι θέλετε να κάνετε κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη στη διαθεσμική συμφωνία για να μπορέσει να συμβάλλει περισσότερο στις διαβουλεύσεις με την Κολομβία ή με, για άλλα εμπορικά θέματα. Δεύτερον, σχετικά με τη συμφωνία Άκτα Πρόκειται ε, ε, για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και φοβόμαστε ότι ε, τα αποτελέσματα του πακέτου τηλεπικοινωνιών που διαπραγματευθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσο αναφορά την προστασία του διαδικτύου θα περιορίσουμε την ε, ελευθερία του. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι δεν ξεπεράσετε ε, τα συμπεφωνημένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα άκτα. Υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε πρώτες ύλες, διότι ορισμένα κράτη ε, στην, στον κόσμο κάνουν, κάνουν ε, πολλά και, και διάφορα και δεν συμφωνώ αλλά ε, θα πρέπει να υπάρχει μία δίκαια εξασφάλιση των πρώτων υλών και εσείς τι πρωτοβουλία σκοπεύετε να πάρετε προς αυτή την κατεύθυνση Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ έχετε πάλι το λόγο για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Πολλέ είναι πάλι ερωτήσεις, έχετε τον ίδιο χρόνο με πριν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω αυτό τι απαντήσει στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων απαντώντας πρώτα απ' όλα σε μία ερώτηση που είχα ξεχάσει από τον πρώτο γύρο εκ μέρου του κυρίου Σόλτ που αφορούσε τον Καναδά. Ήθελα να πω ότι η Ισπανία είναι ένθερμη υποστηρίκτεια της πρόθεσης αυτών των διαπραγματεύσεων, διότι πρόκειται για την πρώτη εμπορική συμφωνία που θα κάνουμε με μια ανεπτυγμένη χώρα και θα έχουμε νέες δυνατότητες εμπορικών αγορών και δίδονται εδώ και μεγάλη σημασία στον τομέα των υπηρεσιών, των κρατικών προμηθειών και των ε, επενδύσεων. Βεβαίως εδώ υπάρχει και η ε, γεωργική ε, η γεωγραφική προέλευση καθώς και το θέμα της ε, εγγύησης ε, άλλων δικαιωμάτων που προσέχουμε ιδιαίτερα. Όσον αφορά το σχόλιο που έκανε ο κύριος Γκάσπαρη για την εμπορική πολιτική πρόθεσμα αναφέρθηκα, ίσως δεν είχα πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσω να το διευκρίσω και δέκα τη παρέμβασή μου, δεδομένου ότι έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Αναφέρθηκα προηγουμένω στη μελλοντική στρατηγική 2020 και για την εξωτερική της διάσταση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η, η εξωτερική διάσταση της ανταγωνιστικότητας να συμπεριληφθεί η στρατηγική 2020, να ενισχυθεί, να προωθηθεί για την πρόθεση αγορές και να μπορέσουν να πέσουν οι φραγμοί μέσω της στρατηγικής εταιρική σχέση μεταξύ ιδιωτικού τομέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μερών. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε για να ανοίξουν αγορέ κρατικών προμηθειών, ε, βιομηχανία και πνευματικής ιδιοκτησίας και να μπορέσουν ε, όλα αυτά τα θέματα να αποτελέσουν ε, μια συμφωνία πλαίσιο. Καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπω έλεγα προηγουμένω, μετά από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα και λογικά θα πρέπει να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τα σχόλιά σα και τι θέσει σα πριν από την αιρινή Σύνοδο Κορυφής. Και υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να κάνω και μία, ένα σχόλιο στην ερώτηση που έκανε ο κύριος Λάγκε σε σχέση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, συζητήσεις για την εμπορική πολιτική. Έχει αναλάβει δεσμεύσεις Προεδρή μας ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό, έτσι όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Είμαστε λοιπόν απόλυτα διατεθειμένοι με την Κομισιό να συνεργαστούμε πολύ στενά ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι για την εξέλιξη των, διαπραγμα... εμπορικών διαπραγματεύσεων. Είπα, με ρωτά ο κύριος Μάρτιν ποια είναι η αξιολόγηση που γίνεται σε στα πλαίσια του Διατλαντικού Συμβουλίου. Το ΤΕΚ μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι σύμφωνα με την αξιολόγησή μας δεν έχει καταλήξει στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και θα πρέπει να δούμε για ποιους λόγους επιβραδύνθηκαν οι εργασίες αυτού του Συμβουλίου. Διότι συγχρόνως γινόταν και διαπραγματεύσει στα πλαίσια του γύρου της Ρόντα, υπήρχαν οι εκλογές, υπήρχαν διμερεί διαφορετικά προβλήματα και στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΤΕΚ που έγινε στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Οκτώβριο αποτέλεσε την επαναβεβαίωση της βούλησης των συμβαλωμένων μερών να υλοποιήσουν κάποια θέματα στο επόμενο ΤΕΚ που θα λάβει χώρα ή κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας ή κατά τη διάρκεια της επομένης. Ούτως ή άλλως πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό, το ντοσιέ αυτό με το οποίο θα ασχοληθεί ο νέος επίτροπος θα δώσει την ευκαιρία να ενισχυθεί ε, το θέμα αυτό και να προχωρήσει. Όσον αφορά την πρόσβαση σε πρώτες ύλες που ανέφερε και ο κύριος Λάγκε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική να ενισχυθεί ώστε να υπάρχει ίσης όρης πρόσβαση σε όλες τις ε, πρώτες ε, ύλες και να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία της Ευρώπης. Μας ε, απασχολεί η μεγάλη μας εξάρτηση από πρώτε ύλες και ήμι κατασκευασμένες ύλες, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει εμείς να ενισχύσουμε την βιομηχανία πρώτων υλών από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχει ασφαλείς προμήθειες πρώτων υλών και σε λογικές τιμές. Το θέμα της Κολομβίας. Πιστεύω ότι οι στόχοι που ακολουθούμε κύριε Μαρτίν είναι οι ίδιοι. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο που κάνατε και τον τόνο της παρέμβασής σας, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα εστίασης του όλου θέματος και όχι ε, θέμα στόχων. Η τελική στόχη είναι κοινή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε οδούς κατανόησης και συνεργασίες για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Εμείς πιστεύουμε ότι ο δρόμος, όπως σας είπα, ο... Η eh, περίληψη είναι καλύτερος από αυτόν του, του... του αποκλεισμού. Και θέλουμε να υπάρχει και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής ώστε να μπορέσουμε τέτοιου είδους αρχές να τις προωθήσουμε. Και αναφέρουμε κυρίως στο θέμα της ε, αηφόρου ανάπτυξης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά το να αποκλείσουμε διάφορους ή να σταματήσουμε τις διαπραγματεύσεις δεν θα βοηθήσει, θα φέρει μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Και όπως σας είπα κύριε Μορέιρα, η κυρία Φερνάντες, αντιπρόεδρος της Ισπανικής Κυβέρνησης, είναι στη διάθεσή σας για να έλθει εδώ και να συζητήσει μαζί σας όσες φορές, όποτε θέλετε, το θέμα της Κολομβίας για να μπορέσει να σας εκθέσει τις απόψεις μας. Το Α400M πρόκειται για διαπραγμάτευση για την ε, κατανομή της αύξησης του κόστους με την ανάδοχο εταιρεία είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται όχι το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Άμυνας. Ελπίζουμε ότι επειδή πρόκειται για ένα σχέδιο πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία επωφελή για όλους. όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Όλες οι απόψεις και οι ανησυχίες που έχετε εκφράσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς στην Επιτροπή σας λαμβάνονται υπόψη στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μας λοιπόν λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία λέτε, αλλά για κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Για θέματα τα οποία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών ή συναρμοδιότητας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά για θέματα τα οποία εξαρτώνται από εμά να είστε σίγουροι ότι δεν θα φυστούμε προσπαθειών για να καταλήξουμε σε αιωνία Επίση είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει ακόμη κανένα κεφάλαιο. Συνεχίζουμε λοιπόν στη γραμμή ότι δεν θα καταλήξουμε σε καμία συμφωνία αν δεν συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία. Δεν ξέρω αν άφησα έξω κανένα σημείο. Όταν μιλούμε για στα πλαίσια του γύρου της Δόχα για συμφωνία φιλόδοξη και σφαιρική μιλούμε για συμφωνία η οποία θα είναι εποφελής και για μας και για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς εμπορικές αγορές και αυτό είναι ο στόχος μας στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα. Επίσης, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ θέλουμε πάντα να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των μελών. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ξεπέρασα το χρόνο που μου είχατε δώσει. Ελπίζω να απέντησα σε όλα τα ερωτήματα. Εάν κάποιος δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις μου, ε, θα επανέλθω αν θέλει κάποιος ή γραπτός ή κάποια επόμενη φορά. Θα σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και εσείς και τα μέλη της Επιτροπής και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος. Εξαιρετική ευκαιρία να ακούσουμε τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας για την εμπορική πολιτική. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας είμαστε γνώμονες για την ε, προθυμία σας να συνεργαστείτε με τα μέλη της Επιτροπής μας. Και την επόμενη φορά, ίσως απλώς να έχουμε πιο συγκεκριμένη συζήτηση με στόχευση σε συγκεκριμένα θέματα. Ο κ. Σεφτάντο Μπονέ που είναι Γενικός Γραμματέας των θεμάτων εξωτερικού εμπορίου και μέλος της, Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής για τις Εμπορικές Σχέσεις του Συμβουλίου. Και εκείνος πρόθυμα συνεργάστηκε μαζί μας. Ευχόμαι λοιπόν στην Ισπανική Προεδρία καλή τύχη για να επιδιώξει και να επιτύχει όσου περισσότερου στόχου τη μπορεί για την Ευρώπη και τι σχέσει τη, τι εμπορικέ γενικότερα. Ευχαριστούμε. attention, please. Time's running. Κυρίες και κύριοι, τρέχει ο χρόνος. Πρέπει να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, προσοχή. Έχουμε μεταθέσει το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης και αυτό θα δούμε. Το εμπόριο και οι οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή μα τον κύριο Μετίν Καζάκ, από την ομάδα Άλντε, που είναι υπεύθυνο για το σημείο αυτό, για την έκθεση αυτή. Το θέμα αυτό δεν το είχε εξετάσει η Επιτροπή μας στην προηγούμενη θητεία, οπότε επήγει να δούμε τις εμπορικές μας σχέσεις με ένα τόσο σημαντικό εταίρο και είναι και το αντικείμενο έκθεσης ιδίας πρωτοβουλία. Συνάδελφοι σας παρακαλώ, πάυσετε, πάυσετε τις διμερείς. On this floor, please. As I was saying, our economic... Όπως έλεγα, οι οικονομικές μας σχέσεις με την Τουρκία είναι ιδιαίτερες. Μιλάμε εδώ για μια χώρα υποψήφια για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Τουρκία είναι και μια από τις λίγες χώρες με τις οποίες έχουμε τελωνιακή ένωση. Πολύ καλές λοιπόν οι σχέσεις μας συνολικά με την Τουρκία, ωστόσο αληθεύει επίσης ότι υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα από εμπορική άποψη και μάλιστα σημαντικά, όπως τα IPR τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, όπου χρειάζεται στενότερη συνεργασία για να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Δίνω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μα για τέσσερα λεπτά και μετά θα προχωρήσουμε στη συζήτησή μας. Κύριε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν ε, αναφέρατε, κύριε Μορέιρα, κύριε Πρόεδρε, τι ιδιαίτερε οικονομικέ και εμπορικέ σχέσει μα με την Τουρκία, πολύ σωστά είπατε ότι είναι ζωτική σημασία. Η Τουρκία είναι ο έβδομο εμπορικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο όγκο των διμερών εμπορικών μα σχέσεων ανέρχεται σε περισσότερο από 100 δι ευρώ. Η Τουρκία είναι ο πέμπτο προορισμό των εξαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει γίνει ο έβδομο παρέχων ε, αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009. Κατά τις ε, χρονιές 2008 και 2009, ο όγκος του εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης γνώρισε μια σχετική ύφεση, ε, εν μέρη λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ε, μειωμένης ζήτησης της Ευρώπης για το τουρκικά εμπορεύματα. Ωστόσο, οι στατιστικέ δείχνουν ότι το 42% του όγκου του εξωτερικού εμπορίου τη Τουρκία κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τι βασικότερε πηγέ για τι ξένε επενδύσει, τι άμεσε ξένε επενδύσει στην Τουρκία. Οι ροέ ε, των ξένων επενδύσεων ε, με προορισμό την Τουρκία έχουν ε, αυξηθεί ιδιαίτερα το 2009, 88% το 2009 σε σχέση με το 5% το 2008. Στόχο μου σε αυτή την έκθεση, Πρόεδρε, είναι να παρουσιάσω μια αποτίμηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με αυτό το σημαντικό εμπορικό μα εταίρο που είναι ένας εταίρος παραδοσιακός, με αλλά βρίσκεται και γεωγραφικά πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ, πολύ άριθμο εμπορικό δυνα... εργατικό δυναμικό, που έχει και πολλά προσόντα και διευκολύνει τι ε, εμπορικέ συναλλαγέ ε, που θα ωφελήσουν ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία την ίδια. Ε, δεν θέλω να σταθώ σε τρει προβληματισμού που αφορούν τι οικονομικέ και εμπορικέ μα σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία και αυτό κατά την εισαγωγή μου. Η πρώτη είναι η Τελωνιακή Ένωση, έπειτα η μη δεσμολογική και μετά η περιφερειακή συνεργασία. Κατά πρώτον, η Τουρκία, όπω το είπατε κύριε Πρόεδρε, είναι η μόνη χώρα εκτό τη Αντόρα και του Σαν Μαρίνο με τι οποίε έχουμε τελωνιακή ένωση ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένωση αυτή ισχύει από το 1996 και τα θεμέλια της ε, βρίσκονται στο πρωτόκολλο της Άγκυρας το 1963. Η Τουρκία, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εποφελείται από τα πλεονεκτήματα αυτής της Τελωνιακή Ένωσης, όμως αυτή η ένωση δεν είναι βεβαίω ακόμη ιδανική. Υπάρχουν διάφορες δυσκολίες. Λόγω χάρη, οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών δημιουργούν μεγάλες ε, δυσκολίες και για τα δύο μέρη, τι δύο πλευρέ, γιατί η Τουρκία δεν είναι ακόμη μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν μπορεί να δεσμευτεί για, και να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσει για συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με τρίτε χώρε. Έχει όμω την υποχρέωση να εγκρίνει τι ίδιε συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτε. που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει με τρίτε χώρε, εφόσον αυτέ έχουν υπογραφεί. Επίση, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει μηχανισμού για να διασφαλίσει την υπογραφή των συμφωνιών αυτών μεταξύ των ε, τρίτων χωρών και τη Τουρκία. Εδώ ήθελα λοιπόν να προτείνω κάποιες συστάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και την αμοιβαία αρρωγή, για το μηχανισμό της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την επίλυση διαφορών. Μετά από πολυάριθμες συναντήσεις και επαφές με την Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Ευρωπαϊκή Επιτροπή της, Μη κυβερνητικέ οργανώσεις Ευρώπης και Τουρκίας, και τους ακαδημαϊκούς ε, και των δύο περιοχών έχω πιστεί ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να λυθούν εκτός πολιτικού περιβάλλοντος. Έπειτα, οι τεχνικοί φραγμοί έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα λόγω των οικονομικών απολειών και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Τουρκία. οι κύκλοι των Ευρωπαίων επιχειρηματιών αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των μέτρων διαφύλαξης, των μέτρων κατά του ντάμπινγκ, των κρατικών βοηθειών, των επιδοτήσεων και το καθεξής. Όλες αυτές οι δυσκολίες είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων και πρέπει να καταλήξουμε σε κοινέ συστάσεις ώστε να καταλήξουμε και σε κοινέ λύσεις για να θεραπεύσουμε αυτά τα προβλήματα. Τέλος, Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό. Η Τουρκία είναι ένας εταίρο ε, καθοριστικός ε, για τον εύξηνο πόντο, την Κεντρική Ασία, τον Κάφκασο, την Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Η εμπορική, πολιτιστική, ιστορική δεσμοί με τις χώρες της γεωγραφικής ζώνης αυτής είναι καθοριστική σημασία και για τη συνεργασία τη δική μας με τις χώρες αυτές γιατί μπορεί να ωφελήσει και τις δύο πλευρές η ευρύτερη αυτή συνεργασία σε ένα πλαίσιο που να έχει πλεονεκτήματα και για τους μεν και για τους δε. Για να ακούσουμε τώρα την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λόγο έχει ο κύριος Άλφερον Τσαλόνε. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως θα θυμάστε, και ο κύριος Καζάκ πολύ σωστά το ανέφερε, η Τουρκία όχι μόνο είναι υποψήφια χώρα για ένταξη, και αυτό βεβαίως δημιουργεί ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εμπορικές αυτές σχέσεις έχουν προωθηθεί χάρη στην Τελωνιακή Ένωση που είναι μοναδική στο είδος της. Είναι πραγματικά μοναδική και λόγω της σημασίας της και σε σχέση με τις άλλες Τελωνιακές Ενώσεις που έχουμε. Τις δύο άλλες δηλαδή, με τα άλλα δύο κράτη. Εδώ δημιουργούνται πραγματικά μοναδικές εμπορικές σχέσεις. Δεν θα θυμίζω τώρα τους αριθμούς που αναφέρθηκαν και με τους οποίους συμφωνώ. Είναι τεράστια σημασία σε εμπορικές σχέσεις για τις δύο πλευρές. Απλώς πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εμπορικός εταίρος της ε, Τουρκίας και αυτό μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Το εμπόριο λοιπόν μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια με μια μικρή ύφεση το 2009 λόγω της ε, γενικότερη χρηματοπιστωτική κρίσης. Εξωγενείς παράγοντες δηλαδή. Όμως η τάση είναι αυξητική. Όλα τα τελευταία χρόνια. Όπως επίσης αναφέρθηκε, Οι εμπορικές αυτές σχέσεις φυσιολογικά δημιουργούν και κάποια προβλήματα, τριγμούς και δυσκολίες. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που είναι εξαιρετικά για αυτές τις, ιδιαίτερα μάλλον για αυτές τις εμπορικές σχέσεις. Οι διαφορές δεν επιλύονται ποτέ μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πλευρών. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρεθεί ένα μηχανισμό επίλυση των διαφορών. Θα μα ενδιαφέραν λοιπόν ε, ιδιαίτερω τα πορίσματα τη έκθεσή σα και τα συμπεράσματά τη και ανυπομονούμε να τα λάβουμε. Μπορεί πραγματικά να καταλήξουμε έτσι σε ένα σημαντικό εργαλείο για να βελτιώσουμε τι εμπορικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Βεβαίω, παραμένουμε στη διάθεσή σα για να συνεισφέρουμε κι εμεί ε, με τη γνώση που μπορεί να διαθέτουμε και εφόσον μας ζητηθεί στην ερευνά σας. Και ευχαρίστως να ξανασυμμετάσχουμε και στη συζήτησή σας εφόσον ετοιμαστεί η έκθεση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα κλείσω εδώ. Okay, thank you. I didn't ευχαριστώ. Ε, δεν σας διέκοψα γιατί θεώρησα ότι δύο λεπτά ίσως δεν επαρκούσαν. για τη συζήτηση αυτή. Δίνω τώρα το λόγο εις ε, τους σκιώδης εισηγητές. Ξεκινάω με τους ε, ε, με το ΕΛΚ όπου η συνάδελφος αποσιάζει Τσέσκο Μπαζάνη Νομίζω ότι ο, μόνο, μόνο ο κύριος Ρόμπερτ Στέρντ είναι εδώ. Ευχαριστώ. Ε, κάποια στιγμή φτάνει και η σειρά μου. Πρέπει να θυμάστε την έκθεση αυτή η οποία αναφέρεται στις οικονομικές σχέσεις και δεν έχει καμία σχέση με ε, την ε, αίτηση για προσχώρηση της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει ήδη μία ασθενή ε, συνεργασία. Καλύπτουμε τις μισές εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε... Η, η Τουρκία είναι η έβδομη χώρα χώρα των ε, δικών μας εξαγωγών. Ε, το 1995 νομίζω είχαμε υπογράψει την εμπορική συμφωνία, την είχα στηρίξει στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα να συνεχίσω να στηρίζω τις εμπορικές σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό χαίρομαι για την έκθεση και το ε, ε, αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν όμως ακούω για τη γεωργία και παρόλο που είμαι γεωργός τρομάζω διότι όταν μιλάει κανείς για γεωργία όλα καταραίουν ταχύτατα. Γι' αυτό το λόγο πάντοτε ανησυχώ και θα ήθελα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Όσον αφορά την εμπλοκή της στη Euromed είναι βασικό η Τουρκία να συμφωνήσει με τους άλλους ε, ομολόγους της στην Euromed και θα ήθελα να ευθυγραμμιστεί περισσότερο στη, ε, ε, στη γραμμή των άλλων χωρών της Euromed προτού προχωρήσουμε περαιτέρω. Νομίζω ότι εδώ θα μείνω. Υπάρχει άλλη ομάδα η οποία θέλει να τοποθετηθεί από αυτού. Κύριος Χίγκιντς, χωρίς μικρόφωνο. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι σε κάθε συζήτηση για τις εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία πρέπει να υπενθυμίσω στην ε, Επιτροπή ότι έχουμε μόνιμες ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών και τη στάση ε, της ε, τουρκικής κυβέρνησης σχετικά με τα θέματα αυτά. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα τα θέματα αυτά δεν είναι κάτι που πρέπει να ξεχνάμε ε, όταν συζητάμε περί εμπορίου. Υπάρχουν τα δικαιώματα των Κούρδων ε, υπάρχει το πρόβλημα της γλώσσας τους, της μειονότητές τους, τα άλλα ε, δικαιώματά τους, αλλά επίσης και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστών στην Τουρκία, επί του οποίου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Η τουρκική κυβέρνηση ούτως ή άλλως ακολουθεί την ίδια ε, πολιτική φιλελευθερισμού που ακολουθούν και περισσότερες κυβερνήσεις Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, όταν, όσον αφορά την επιχείρηση ΤΕΚΕΛ η οποία λέγεται ότι ε, θα ιδιωτικοποιηθεί και που απεργούν οι εργαζόμενοι εδώ και 43 ημέρες γιατί προβλέπεται θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Εξ αυτών 40 αυτή τη στιγμή κάνουν απεργία πίνης και ε, η χώρα, η, από, η επιχείρηση αυτή έχει το μονοπόλιο των προϊόντων καπνού και υνοπνευματοδών ε, και πρέπει να πω ότι θα πρέπει να κόσουμε τους εργαζομένους στην Τουρκία επί του συγκεκριμένου θέματος προτού αποφασίσουμε. Ο Λόρδος Ντάρτμουρθ από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Στέρντι ε, πολύ ε, χλιαρά στήριξε την Τουρκία διότι είπε ότι στηρίζει την ε, εμπορική συμφωνία διότι η το κόμμα το οποίο τόσο επάξια εκπροσωπεί ο κύριος Στέρντι ε, στηρίζει πλήρως την Τουρκία και την πρόοδό της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έπρεπε να το έχει τονίσει πίσω ο κύριος Στρόερντι. Εάν λοιπόν έχουμε τόσο στενή θέση, ε, σχέση με την Τουρκία, αν το ίμιση των εξαγωγών της Τουρκίας έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να συμμετέχουν συμμετέχει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κανένα βία ή κάποιο σοβαρό λόγο να γίνει μέλος Ευρωπαϊκής Ένωση. και εφόσον υπάρχουν σημαντικά θέματα δημοκρατικά και ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία ε, θα πρέπει ε, να έχουν εκπληρωθεί προτού εξετάσουμε ε, την πρόοδο της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να λάβουμε υπόψη ε, την ε, προσχώρηση 70 εκατομμυρίων εργαζομένων με ε, ένα κατακεφαλήν εισόδημα που είναι το μισό από αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα δύο λεφτά για να σχολιάσει τη θέση την οποία εξέφρασαν οι διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο, διότι δεν νομίζω ότι είναι ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει στο πεδίο και στο περιεχόμενο μια έκθεση που ούτω ή άλλω είναι έκθεση ιδία πρωτοβουλία. Θα περνάγαμε σε θέματα που ξεπερνούν το εμπορικό πεδίο. Προτιμώ λοιπόν να μην προσθέσω σχόλια σε αυτά. Uh, και τελευταίο σχόλιο από τον εισηγητή μας, κύριε Καζάκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ευαισθησία... Δύο λεπτά, μάλιστα. Η ευαισθησία, λοιπόν, τη συζήτηση αυτή για τα θέματα της Τουρκίας είναι κατανοητή. Αλλά να θυμίσω ότι ήδη Υπάρχει ετήσια έκθεση περί Τουρκίας, η οποία συζητήθηκε στο επίπεδο της ε, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής μάλλον Εξωτερικών Υποθέσεων και όλα τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα πολιτικά ζητήματα συζητήθηκαν για μακρόν. Σκοπός της έκθεσής μου στην δική μας την Επιτροπή του Εξωτερικού Βορείου είναι να δούμε τις εμπορικές σχέσεις μας μόνο υπό το πρίσμα το αυστηρός οικονομικό και εμπορικό Δηλαδή, πώ μπορούν οι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία να αναθερμανθούν, να προωθηθούν. Από τεχνική άποψη, τι χρειάζεται για τη συνεργασία μα. Τι προσέγγιση πρέπει να καταρτήσουμε ώστε να έχουμε πλεονεκτήματα και για του μεν και για του δε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όλε οι διαπραγματεύσει σε σχέση με την ε, πορεία της προ την ένταξη δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο για τι οικονομικέ και εμπορικέ μα σχέσει ούτως ή άλλως. Αυτό λοιπόν θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους, να μην ξεχάσουν αυτήν την οπτική για το θέμα και αυτή την προσέγγιση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα συζητήσουμε το θέμα το Μάρτιο, δημόσια ακρόαση. Εξέταση τη έκθεση στην Επιτροπή τον Απρίλιο, κατάθεση για, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών τον Μάιο. Εξέταση των τροπολογιών αρχίζει τον Ιούνιο και θα ψηφιστεί η έκθεση στην Επιτροπή μα τον Ιούνιο του 2010. Πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Να πάμε πίσω τώρα στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα GSP SIN στην Κολομβία. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με αρκετούς προσκεκλημένους που έχουν επιλεγεί από τους συντονιστές εδώ έχουν δοθεί προτιμησιακές, ε, έχουν προβλεφθεί προτιμησιακά μέτρα σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και αυτά στα πλαίσια του προγράμματος GSP SIN. Αυτό το πρόγραμμα για την αναπτυγμένη περιφερειακή εμπορική συνεργασία προτείνει δασμολογικές προτιμήσεις με τη μείωση ή και την εξάλληψη εισαγωγικών δασμών για τις ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες όμως κυρώνουν και υλοποιούν τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, ιδίως σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακών δικαιωμάτων, βιώσιμης ανάπτυξης και καλής διακυβέρνησης. Υπάρχουν ειδικέ διευθετήσει που απαιτούν από τι χώρε αυτέ να καλύπτουν πολλέ προποθέσει. Πρώτα απ' όλα να έχουν κυρώσει και ενεργώ υλοποιήσει όλες τι συμβάσει που απαριθμώνται στο παράρτημα 3 του προγράμματο GSP. Έπειτα να αναλάβουν την κύρωση των συμβάσεων και να προβλέψουν στην νομοθεσία τους μέτρα ώστε να παρακολουθούνται και να ελέγχονται τα επιτεύγματα της υλοποίησης. Ανάλογα με τα όσα προβλέπονται για τις απαραίτητες χώρες. Ο κανονισμός προβλέπει προσωρινή απόσυρση κάποιων εκτιμάτων του προγράμματος εάν η εθνική νομοθεσία δεν αντικατοπτρίζει τις απαιτήσει των διεθνών συμβάσεων ή εάν δεν απο... υλοποιείται αποτελεσματικά. Οι διάφορε οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συνδικαλιστικέ οργανώσεις έχουν εκφράσει ανησυχίε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία συγκεκριμένα. ιδίω ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων και τι δράσει των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η Επιτροπή μα λοιπόν αποφάσισε να οργανώσει ανταλλαγή απόψεων για το πρόγραμμα GSPC και την υλοποίησή του στην Κολομβία με τον πρέσβη τη Κολομβία και εκπροσώπου των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό με τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα και τι νέε ευθύνε του Ευρωκοινοβουλίου για τα εμπορικά ζητήματα, πρέπει να δούμε κατά πόσον η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται και το πρόγραμμα GSPC πρέπει να άρει τα ωφελήματά του για την Κολομβία. Η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο λοιπόν ενδιαφέρονται ιδιαίτερως να παρακολουθήσουν το πώς γίνονται αντιληπτά τα ωφέλη του προγράμματος αυτό από τις δικαιούχες χώρες. Είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε μαζί μας σήμερα μερικού επαΐοντες για το θέμα αυτό με ιδιαίτερη πείρα στον τομέα τους, οι οποίοι μπορεί να μας διαφωτίσουν και να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεών μας και την κατανόηση της, της κατάστασης στην Κολομβία για μας ώστε να έχουμε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον κύριο Αλμπέιρο Φαλτεράμα, ο οποίος είναι πρόεδρος του τμήματος της για τις, αγρο... για τις γεωργικές δραστηριότητες ανάπτυξης. Ε, ακολουθεί ο κύριος Βανέγκας, ο οποίος εκπροσωπεί το Κεντρικό Συνδικαλιστικό Όργανο Εργαζομένων και αυτοί είναι οι βασικοί μας ομιλητές. Θα δώσω το λόγο σε καθέναν με τη σειρά, ξεκινώντας από τον κύριο Φράνκο Βαλτεράμα 8 με 10 λεπτά το πολύ ο καθένας. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Ευχαριστούμε που ήρθατε για να συμμετάσχετε σε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση. Κύριε Ερίκε Φράνκο Βαλτερά, έχετε το λόγο. Γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που μας δίδει την δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούγεται στη, στη χώρα μου. Εγώ εκπροσωπώ έναν τομέα στη χώρα μου τις μπανάνες, την ε, οικοδομή, την ε, ανθοκομία και ένα μεγάλο συνδικάτο γενικότερα με κατασκευαστικές εργασίες. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εμείς είμαστε εδώ ως εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων και αρχίζοντας θα πω ότι πιστεύουμε ότι κάποια μειονοτικά συνδικάτα πρέπει να μείνουν εξ ονόματο του και όχι εξ ονόματο όλη τη της ε, τη Κολομβία. Τελευταίε εκλογέ το 2006, ένα μειονοτικός ε, τομέα του δικού μα ε, κοινοβουλίου ζήτησε να ψηφίσουμε κατά όλων αυτών που ήθελαν να προχωρήσει η εμπορική συμφωνία με τη Αυτό ήταν μεγάλη ήττα, δεδομένου ότι με πολύ συντριπτική πλειοψηφία εκ μέρους των κυβερνώντων και της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο μας ψηφίστηκε αυτή η συμφωνία. Οι περισσότεροι λοιπόν ζήτησαν να υπερψηφιστεί και υπερψηφίστηκε αυτή η σύμβαση ελευθέρου εμπορίου με τις, είπα και την ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι σωστό να ζητείτε ε, από την κοινωνία να καταψηφίσει ε, τη συμφωνία αυτή. Επίσης πρέπει να σας πω ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι πάρα πολύ αδύναμο. Υπάρχουν μόνο 4% εκπροσωπούμενοι εργαζόμενοι στο συνδικάτο αυτό. Η... Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο εισέχεται στην τελευταία ολομέλεια του το, 2... 2009 αποφάσισε να συμμετάσχει στην διαδικασία διαπραγματεύσεων και να μην ε, περιοριθεί όπως κάνει η ΚΟΥΤ. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Κολομβίας ψήφισαν υπέρ αυτών των ε, συνθήκων και πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι κάτοικοι της Κολομβίας είναι απλοί εργαζόμενοι και δεν είναι κατά της διαπραγμάτευσης ε, σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, μας απασχολεί το ότι γίνονται προσπάθειες να μην υπάρχει σύστημα ε, πρόνοια στη χώρα μας. Κάτι τέτοιο συμβεί, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους εργαζόμενους στην Κολομβία και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι έχουμε μεγάλα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα, άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το σύστημα μέχρι να μπορέσει να υπογραφεί αυτή η εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνουν ε, οι συνδικαλιστικές ενώσεις σε σχέση με την απόρριψη των συγκηθικών είναι να κάνουν απόρριψη αυτών των συνδικών για λόγους ιδεολογικούς. Εγώ πιστεύω ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να είναι εποφελής ε, για όλα τα συμβαλόμενα μέρη και να μην υπάρχει εκμετάλλευση των αδυνάμων ε, από τους δυνατούς. Μόνο έτσι πρέπει να προχωρήσουμε νομίζω χωρίς να είμαστε δογματικοί και να εγκαταλείπουμε και να ε, απορρίπτουμε τα πάντα πριν να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει να πω ότι στον τομέα αυτό αυτή τη στιγμή που είμαστε σε ε, προεκλογική εκστρατεία διότι έχουμε βουλευτικές ε, εκλογές τον επόμενο μάρτιο, γίνεται προσπάθεια εκ μέρους κάποιων συνδικάτων να απορριφθούν όλες οι συμφωνίες ο το, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αρχίζοντας λέμε ότι δεν υπάρχει ειδικό πρόβλημα ε, γενοκτονίας των εκπροσώπων των συνδικάτων, όπως είπαν κάποιοι. Πρόκειται για μύθο πρέπει να πω ότι όντως είμαστε θύματα βίας εδώ και διάφορες, εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ε, εμείς οι συνδικαλιστές ε, θύματα Επίσης πρέπει να πω ότι σύμφωνα με τις ε, στοιχεία της αστυνομίας δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θύματα μεταξύ μας, αλλά και πάλι όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία δεν μπορούμε πάντα να τα επαληθεύουμε. Πρέπει να πω ότι σήμερα, όπως σας έχω πει, τα τελευταίες, τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί πολύ ο πληθυσμός μας, αλλά πάρα πολύ λίγο η συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα. Δεν μπορώ να πω ότι ε, ο κόσμος είναι ιδιαίτερα βίαιος κατά των συνδικαστικών. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι είμαστε αντίθετοι με αυτούς που επιβεβαιώνουν ότι ο συνδικαλισμός είναι η πιο ε, επικίνδυνη οργάνωση στην Κολομβία. Σύμφωνα με στοιχεία της αγγελίας, Το 2005 στην Κολομβία αποτέλεσαν αντικείμενο επιθέσεων έμποροι, φοιτητέ, νέοι, διάφορα άτομα τα οποία ε, ασκούσαν διάφορα επαγγέλματα Και από τις διάφορες στατιστικές που έχουμε, το να είναι κανείς συνδικαλιστές σημαίνει ότι είναι λιγότερο αντικείμενο βίας παρά από το να ανήκει σε κάποια άλλη επαγγελματική τάξη. Ακόμη ένα λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Ξέρουμε ότι από το 1983 έχουν ε, αποτελέσει, έχουν δολοφονηθεί γύρω στις 2.500 συνδικαλιστές. Αυτό όμως σε σχέση με τα υπόλοιπα άτομα του πληθυσμού δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός ο αριθμός. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε επίσης ότι όταν γίνεται λόγος για συνδικαλιστές που έχουν οριστεί από κάποιους άλλους μιλάμε για όχι σαφή θέση του συνδικαλισμού. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο τον δεύτερο κύριο μιλητή, τον κύριο Αλμπέρτο Βάνεγκας. Διευθυντή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ΚΟΥΤ, Κεντρικό Συνδικάτο της Κολομβίας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και εξ ονόματες της ΚΟΥΤ για την δυνατότητα που μας δίδεται να σας μιλήσουμε για καταστρατηγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των συνεκαλιστών στην Κολομβία. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην πολιτική συζήτηση που θα γίνει για την έγκριση ή όχι Μία ε, συνθήκη ελευθέρου εμπορίου μεταξύ Κολομβίας και, Ηνωμέν... και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν αρχίσω και σεβόμενος πλήρως τους ε, παρόντε θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση όσον αφορά την παρουσία του κυρίου Αλμπέιρο Φράγκο, ο οποίος είναι μέλος της ΣΕΖΕΤΕ, τον οποίο ε, γραπτός στον οποίο αυτός απαγόρεψε το δικό του συνδικάτο να λάβει το λόγο. Άρα ο κύριος Φρανκό μιλά ε, εξ ονόματός του μόνο. Ως ε, συνδικάτο θα πρέπει να εκφράσουμε την ησυχία μας για την πολύ σοβαρή κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ανθρώπικα δικαιώματα και την καταστρατήγηση των ε, συνδικαλιστικών ελευθεριών στην Κολομβία. Είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθεί ένα νέο συνδικάτο ή ακόμη και στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε συλλογικές συμβάσεις ή να απεργήσουμε. Η κατάσταση αυτή είναι η κατασταση αυτη ειναι κατασταση την οποία δαπιστώνει εδώ και ε, δεκαετίες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διεθνής οργάνωση εργασίας και το Ηνωμένα Έθνη. Η Κολομβία ξέρουμε ότι είναι κατεξοχήν η χώρα η οποία καταστρατηγεί τα δικαιώματα των ανθρώπων. Στην τελευταία σύσκεψη τον Μάρτιο του 2009 τη Διεθνής οργάνωση Εργασίας η Κολομβία ήταν στον κατάλογο των 25 κρατών που παραβιάζουν περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε καταρρύπτοντας ε, την ε, θέση της ε, κυβέρνησης που κάνει τρομερές διπλωματικές προσπάθειες για να καθαρίσει την εικόνα την οποία έτσι κάνοντας χειραγωγή στις στατιστικές ενώ τα γεγονότα πολλές φορές για να μην πω συνέχεια τους ενέχουν σε διάφορα ε, θέματα καταστρατήγησης των δικαιωμάτων. Ε, πολλοί είναι φυλακισμένοι διότι συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές όργανων. και νομίζω ότι πολλές φορές άτομα της αντιπολίτευσης από συνδικαλιστές έως και δικαστές βρίσκονται ακόμη στην ε, φυλακή. Ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις όπως στη Σουέτσα νέοι οι οποίοι ε, είχαν ε, κατηγορηθεί ε, ελευθερώθηκαν τελικά μέσα σε ένα πλήρες καθεστώς ατιμορρησίας. Η Κολομβία έχει δραματικό ρέκορ 60% δικαλιστών που έχουν δοφλοφονηθεί στον κόσμο. Κατά την διάρκεια των δύο θητιών του ΡΙΜΠΕ θανατώθηκαν 573 δικαλιστικοί εκπρόσωποι, 39 το 2007 και όλες αυτές οι περιπτώσεις ε, είναι περιπτώσεις στην οποία ο δολοφόνος χαίρει καθεστώτος ελευθερίας και πλήρους ατιμορρησίας. πρέπει να πω ότι πολλές φορές οι αποφάσεις ε, ε, των δικαστηρίων αφορούν ε, ελάσσονος σημασίας παραπτώματα ή αδικήματα, ενώ όπως σας είπα, επαναλαμβάνω, είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δολοφονίες συνδικαλιστών θέματα τα οποία ε, φεύγουν από τα δικαστήρια και μένουν ελεύθεροι και ατιμόρυτοι οι δολοφόνοι. Στον ε, τομέα της εκπαίδευσης πρέπει να πω ότι δολοφονείται κάθε εβδομάδα ένας εκπαιδευτής εδώ και πέντε χρόνια τουλάχιστον. Και εμείς ε, καταγγείλαμε εθνικός και διεθνώς την ευθύνη του κράτους της Κολομβίας που είναι θετικά ή αρνητικά υπεύθυνο τα πιστηματα Η κυβέρνηση όμως πρέπει να σας πω ότι πάντα παρουσιάζεται ως θύμα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απεδείχθη ότι πρόκειται για πράκτορες του κράτους. Ε, αυτοί είναι οι οποίοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην περίπτωση τριών συνδικαλιστών της Ραούκα το 2006 πρέπει να σας πω ότι ο Φραγκισίσκο Σάντος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παρουσίασε ε, ε, την περίπτωση αυτών των τριών ότι πέθαναν στον χώρο της εργασίας τους, ενώ ξέρουμε εκ των υστέρων ότι δολοφονήθηκαν. Υπάρχουν τρία συνδικαλιστικά όργανα και διάφορες οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών και όλοι μας έχουμε πει να μην υπογραφεί αυτή η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κολομβίας αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων καθώς και άλλοι διεθνείς οργανισμοί μας υποστηρίζουν και αυτή η ανθρωπιστική κρίση στην οποία βρισκόμαστε και μέσα στην οποία προσπαθούμε να αναπτύξουμε το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ήδη έχουν συναυθεί συμφωνίες με τις είπαμε με τον Καναδά και πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να ακρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για να μην βρεθεί σε τέτοια αμφιλεγόμενη κατάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό εξάλλου προβλέπεται και στην ε, ε ιδρυτική της συμφωνία. Πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορες ρήτρες ανθρωπιστικού περιεχομένου τις οποίες έχει ε, παραγνωρίσει η δική μας κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι θέλησε προς το παρόν να αναβάλει την εφαρμογή του ΣΕΧΕ ΣΥΝ ώστε η Κολομβία να μπορέσει να συμμορφωθεί. Γι' αυτό ζητούμε να παθό να ανασταλεί η εφαρμογή του ΣΕΧΕΣΕ ΣΥΝ και δεύτερον να σταματήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω διαπραγμάτευση για την υπογραφή της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου με την Κολομβία. Είμαστε πεπισμένοι, εμείς οι εργαζόμενοι, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι μια αξία την οποία θα πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας και σας ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. This, uh, now we Ευχαριστούμε. Και τώρα θα τοποθετηθούν ε, Ακούσαμε μάλλον τις απόψεις των δύο πλευρών που όπως αναμενόταν ήταν διαφορετικές. Και τώρα οι συνάδελφοι θα πάρουν το λόγο για να τοποθετηθούν. Ο κύριος Κάλλος Τροχίλιο για να μας εκθέσει τις απόψει του πρέσβη τη Κολομβία παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι λεπτά το πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμό σε εσάς, καθώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής σας και στους επισκέψεις σας και να επαναλάβω τις ευχαριστίες της χώρας μου για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση που επικρατεί στην Κολομβία. Θα ήθελα επισήμως να ζητήσω από την Προεδρία παρακαλώ να γνωρίσετε σε όλα τα μέλη να, διανύμετε σε όλα τα μέλη του, της Επιτροπής σας τα κείμενα στα οποία φαίνεται από τις στατιστικές πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην χώρα μου για να μπορέσουν να σε ενδιαφέρει τη δουλειά στην Κολομβία να ενημερωθούν καλύτερα. Απ' την άλλη κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να πω στην Επιτροπή σας που ασχολείται με θέματα που αφορούν το εμπόριο, ότι η Κολομβία είναι μία χώρα φίλη του εμπορίου. Είναι μία χώρα φίλη του ανοίγματο των οικονομικών της συνόρων. Είναι υπέρ της σύναψης εμπορικών συμφωνιών με τις ε, ε, διαφορούς διεθνείς ανά τον κόσμο. Είναι υπέρ της ε, σύναψης συμφωνιών για τις ε, προεδρίες είναι κατά της, υπέρ της κατάργησης της διπλής φορολόγησης και είναι υπέρ οικονομικών και εμπορικών συμφωνιών που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της κατάστασης, στη δημιουργία νέων ευκαιριών, θα δημιουργήσουν ε, ε, ένα σύστημα προστασίας κατά της βίας. Απ' την άλλη θα πρέπει να πω ότι η Κολομβία θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για το SHP του οποίου η αναγνώριση το, οποίο η ουσία είναι η αναγνώριση της ε, ε μεγάλης μάχης που κάνουμε κατά των ναρκωτικών ουσιών. Θα ήθελα να κάνω έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υποφελούμε σε ευκαιρίες που είμαι εδώ για να συνεχίσουμε να προχωρούμε από κοινού για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το παγκόσμιο πρόβλημα των ναρκωτικών λέγοντας ότι οποιαδήποτε ε, πράξη συνεργασίας με την Κολομβία σημαίνει επίσης και βελτίωση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι παγκόσμια, είναι οικουμενική, κάτι το οποίο συμμερίζεται και η κοινωνία της Κολομβίας και το κράτος και η κυβέρνηση. Γι' αυτό η Κολομβία πρέπει να πω ότι είναι μια ανοιχτή χώρα σε οποιαδήποτε έλεγχο ή εποπτεία διεθνής. Γι' αυτό όλες οι οργανώσεις, που ανήκουν στα Ηνωμένα Έθνη είναι παρούσες στην Κολομβία. Αναγνωρίζουμε επίσης την νομιμότητα και την αρμοδιότητα της ε, Διαμερικανικής Επιτροπής Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είμαστε πάρα πολύ ενεργοί όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια του ΟΗΕ και πρέπει να πω ότι εφελουσίως έχουμε ε, τεθεί στη διάσκεψη και όλων των εποπτικών οργάνων του ΟΗΕ όσον αφορά την ε, συμμόρφωσή μας και τη δέσμευσή μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα χρόνο μετά ε, παρουσιάσαμε σχετική αναφορά εθελουσίας όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ειδικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον ΟΗΕ. Η βία στην Κολομβία μας απασχολεί περισσότερο από τον καθένα, δεδομένου ότι πρόκειται για τη χώρα μας και αυτοί οι οποίοι δολοφονούνται είναι συμπολίτε μας. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες να ξεπεράσουμε τη βία και έχουμε την ε, διασφάλισε ότι η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολοβία εξαρτάται από το εάν θα κατορθώσουμε να βάλουμε φρένο, αν μπορέσουμε να σταματήσουμε την ε, βία. Και αυτού του είδους οι συνθήκες θα μας βοηθήσουν να το κατορθώσουμε αυτό. Δεδομένου ότι μέσω αυτών των συμβάσεων γίνονται νέες επενδύσεις, δίδονται νέες ευκαιρίες, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης ε, βγάζουμε πολλούς Κολομβιανούς από την παραοικονομία και το παράνομο εμπόριο των ναρκωτικών και έτσι ελπίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα κλίμα ειρήνης και ε, ηρεμίας, πράγμα που θα συνεισφέρει και στην καλύτερη πράξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίως ξέρουμε ότι εδώ υπάρχουν ε, εντελώ αντίθετες απόψει που εκφράστηκαν εδώ, γιατί θα ήθελα επίσημω να σα ζητήσω κύριε Πρόεδρε να θέσετε σε γνώση όλων των μελών τη επιτροπή σα την τελευταία έκθεση της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας την οποία κατήρτισαν οι εμπειρογνώμενες, την οποία υπάρχει ε, ρητή αναγνώριση της βελτίωσης της κατάστασης στην Κολομβία, της μείωσης της βίας γενικά και βεβαίως της μείωσης της βίας ε, κατά των συνδικαλιστών. Τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κολομβιανών υποστηρίζει τις ε, συμφωνίες ελευθέρω εμπορία. Ανεξάρτητες μελέτες αποδεικνύουν ότι όταν ε, γίνεται συμπατριώτες μου αυτή η ερώτηση, το 72% των Κολομβιανών όταν έγινε η σχετική ερώτηση στην Κολομβία, με σαφέστατο τρόπο το 70% του συμπολιτών μου είπαν ότι είναι υπέρ της προσχώρησης σε μια τέτοια συμφωνία. Και νομίζω ότι σεβόμενοι δημοκρατικά και τις απόψεις μειοψηφίας πρέπει να πω ότι αυτό το ποσοστό είναι συντριπτικό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Είναι καλό και σε σχέση με τους προηγούμενους ομιλητές να έχουμε και μια εξωτερική τοποθέτηση. Ο κύριος Ατσεβαρία τώρα από την Εθνική Ένωση Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων Και πάλι έχετε το λόγο για έξι παρακαλώ λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των βιομηχάνων στην Κολομβία αισθάνομαι μεγάλη τιμή που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο λαμβάνω τον λόγο, λαμβάνουμε ως οργάνωση τον λόγο για πρώτη φορά. Οι επιχειρηματίες και οι βιομήχανοι στην Κολομβία σεβόμεθα πλήρως τις διεθνείς συμβάσεις και τα συμβάσεις των ανθρώπινων δικαιώματα. Πρέπει να πω ότι τα τελευταία 15 χρόνια εργαστήκαμε εντατικά για να εξεύρουμε μηχανισμούς ενσωμάτωσης, όχι μόνο στην Κολομβία, αλλά και Διεθνώ ώστε να μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα αυτέ οι συνθήκε. Σε μια χώρα στην οποία υπήρχε στο παρελθόν μεγάλη βία, προσπαθούμε σήμερα να υπάρχει διαφορετικό όραμα και διαφορετική κατεύθυνση. Θέλουμε ε, τους αξίες αυτές να τις μεταφέρουμε και σε άλλες κοινωνίες του κόσμου ώστε οι υπηρεσίες μας, τα προϊόντα μας να αναγνωριστούν ως προϊόντα τα οποία θα διεισδύσουν στις διεθνείς κοινότητες. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι εργασίκαμε σε προγράμματα συνεργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2001 με την υποστήριξη της κυβέρνησης και των εργαζομένων της Σουηδίας έχουμε κάνει ένα διμερές πρόγραμμα με τους εργαζομένους τους ε, στην Κολομβία για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, για την βελτίωση ε, των κοινωνικών σχέσεων. Εγώ είμαι μέλος διαφόρων επιτροπών και μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν τρομερές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Το 2006 κάναμε τριμερή συμφωνία με τους εργαζομένους και τους εργοδότες και την κυβέρνηση όπου τονίσαμε την ανάγκη να βελτιωθεί η δικαιοσύνη ώστε να μην υπάρχει ατιμωρησία όταν έχουμε να κάνουμε με εγκλήματα και κυρίως με εγκλήματα κατά των συνδικαλιστών. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους συνδικαλιστές. Έχουμε δημιουργήσει διάφορες επιτροπές στη χώρα μας ώστε να υπάρχουν ικανοί πόροι για να έχουμε ένα σύστημα προστασίας και βελτίωση ε, των συνθήκων εξερεύνησης των διαφόρων προβλημάτων. Επίσης, ε, έχουμε κάνει προσπάθειες για να αλλάξει η νομοθεσία. Η μάρτυρα των προσπαθειών μας τα τρία τελευταία χρόνια είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ήταν παρούσα, έκανε ε, διάφορες εκθέσεις, η Διευθύντρια, ε, η υπεύθυνη επίσης έκανε μία αφορά ε, μία αναφορά για τη χώρα μας, την οποία τονίζει ότι έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Και πρέπει να πω ότι Στην ε, Σύμβαση 87 έχει δοθεί πολύ καλός βαθμός στην Κολομβία τη συμπεριφορά της. Πρέπει να πω ότι είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ένα κατώτατο μισθό. Και παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, τα τρία συνδικάτα, οι εργοδότες και η κυβέρνηση έχουν κάνει μία κοινή δήλωση, την οποία θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας γνωστοποιήσουμε. Εκεί τονίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε χαμηλό ποσοστό πληθωρισμού. Πέρσι είχαμε 2% τέτοιο ποσοστό πληθωρισμού. Υπογραμμίζουμε την ε, σημασία να γίνει καλύτερο ο κοινωνικός διάλογος, όπου ε, έχουμε ορίσει ημερήσια χρονοδιάγραμμα εργασιών μεταξύ μας για φέτος. Ζητούμε να θεωρηθούν οι πολιτικές της κυβέρνησης της Βενεζουέλας σε σχέση με τις διάφορους περιορισμούς που τίθεται για το εμπόριο με την Κολομβία. Πρέπει να πω ότι ε, οι εμπορικές μας συναλλαγές αυτή τη στιγμή και οι εξαγωγές μας προς την Βενεσουέλα έχουν μπλοκαριστεί, πράγμα το οποίο αποτελεί πρόβλημα και για το λαό μας και για το λαό της Βενεζουέλας. Επίσης πρέπει να πω ότι κάνουμε έκκληση διάφορες διάφορα πολιτικά κόμματα να μην υποστηρίζουν τρομοκρατικές ομάδες. Πρέπει να πω ότι το 50% των εργαζομένων ε, στην Κολομβία δεν βρίσκονται σε κανονικό εργασιακό καθεστώς και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι εμείς από τη μεριά των επιχειρηματιών και βιομηχάνων κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιωθεί η κατάσταση και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το δείτε βάσει διαφόρων δικτών που έχουμε. Επίσης, το 2,7% των εσόδων των μεγάλων επιχειρήσεων πηγαίνουν σε προγράμματα που ξεπερνούν τη δέσμευση που έχουμε επισήμως αναλάβει σε σχέση με αυτά τα οποία ορίζει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προσδίδουμε σε αυτό το θέμα μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί μεγάλη προς, ε, πρόοδος ε, με την ε, εκτέλεση προγραμμάτων βελτίωση των καταστάσεων και πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι συμβάσεις που προβλέπονται θα είναι επωφελείς για όλους. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής, αλλά υπάρχει ένα προβληματάκι, διότι αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μία ώρα σε αυτή τη συζήτηση και όχι περισσότερο. Και έχω τουλάχιστον 7 αγορητές που έχουν ζητήσει το λόγο. Εάν μιλήσετε από 5 λεπτά, Μάλλον από δύο λεπτά θα έχουμε 14 λεπτά. Ε, δεν τον έχουμε τόσο χρόνο. Αποφύγετε λοιπόν τις ερωτήσεις ή τα σχόλια που είναι ίσως περίτα. Θα θέλαμε να ξανακούσουμε τους προσκεκλημένους μας, γι' αυτό να αφήσουμε λίγο χρόνο για να απαντήσουν και στις ερωτήσεις που ε, ο κύριος Θάλμπα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο σύντομο γίνεται. Η κατάσταση στην Κολομβία πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι είναι δύσκολη. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υπάρχει ιδεατή κοινωνία. Άρα θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές και να δούμε πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα. Και πιστεύω ότι οι εξελίξεις από ό,τι βλέπουμε από το 2001 έως τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικές. Όσον αφορά τις δολοφονίες του αμάχου πληθυσμού, ξέρω ότι τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν κατά 45%. Και επίσης, δολοφονίε συνδικαλιστών μειώθηκαν κατά 81%. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι ε, εργάζεται πολύ σωστά κατά της βίας η κυβέρνηση της Κολομβίας. Επίση, θα ήθελα να τονίσω το εξή. Ο ΙΕ θα προτείνει στο Μεξικό να εγκρίνει το πρότυπο της Κολομβίας για την προστασία μη κυβερνητικών οργανώσεων και προστασία του τύπου. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι δεν τα πάει και άσχημα η κυβέρνηση της ε, Κολομβίας από τη στιγμή που το προτείνει στο μεξικό ως μοντέλο ΟΗΕ. Εξάλλου, όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης, η συντριπτική πληροψηφία ε, των Κολομβιανών είναι υπέρ της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Πράγμα το οποίο είναι απόδειξη της δημοκρατίας, εάν θέλει κάποιος να προωθήσει μια τέτοιου είδους συμφωνία. Δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτή τη δυνατότητα από τους Κολομβιανούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όταν ε, συνάπτουμε μία εμπορική συμφωνία με μία άλλη χώρα ή δημιουργούμε ένα θέμα προτιμήσεων ε, τότε ε, είναι μία ανταμοιβή για κάποια εξέλιξη. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε αν βασίζεται όντως σε μία αιτιολογημένη πρόοδο και αν υπάρχει βία η βία αυτή, και η βία αυτή δεν διώκεται πρέπει να ρωτήσω τον πρέσβη ε, γιατί δεν διώκονται οι εγκληματίες ε, εφόσον η δικαιοσύνη είναι μέρος ε, των κρατικών δικαιοδοσιών. Επίσης στο θέμα της βίας υπάρχει μία, ένα σαφής διαχωρισμός των αρχών από αυτούς ε, στους οποίους εξασκείται η βία. Δηλαδή ακούμε ότι εκτός των στρατιωτικών υπάρχουν και παραστρατιωτικές οργανώσεις, ότι υπάρχουν ε, γερουσιαστές και βουλευτές για τους οποίους υπάρχει κατηγορία ότι έχουν σχέσεις με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις και όταν δούμε ε, ότι υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της πολιτικής πολιτικής και αυτών των παραστρατιωτικών οργανώσεων έχω μια μισή, ένα λεπτό μου είπατε. Δεν αντιλαμβάνομαι πόσο διαχωρίζεται η κρατική βία από την ε, ε, ε, το κράτος δικαίου και νόμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθώ να είμαι σύντομη. Θέλω να σας ευχαριστήσω διότι ξεκινήσατε αυτή τη συζήτηση και εξηγήσατε ποιες είναι οι διατάξεις για τα GSPs ε, είμαι νέα ευρωβουλευτήνα και πρέπει ακόμη να ενημερωθώ. Έχω όμως ένα έγγραφο και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει λοιπόν ότι οι αποδέκτες των προτιμησιακών καθεστώτων πρέπει όντως να έχουν εφαρμόσει οι 27 συγκεκριμένες συμβάσεις σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ λοιπόν ε, ε, ε, είμαι προβληματισμένη διότι την περασμένη εβδομάδα κοιτούσαμε τη Σρι Λάνκα όπου υπήρξε κάποια έρευνα και ε, τον ίδιο μήνα που τελείωσε ένας εμφύλιος πόλεμος και τώρα προσπαθούμε ε, να ε, τους αποσύρουμε αυτά τα προσόντα. Οπότε αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δολοφονίες συνδικαλιστών, δασκάλων, αγροτών ή κατά των ε, ηθαγενών και από την άλλη πλευρά άλλοι μας λένε ότι δεν, είναι, δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Πρέπει εδώ να προσπαθήσω να διαμορφώσω ίδια γνώμη. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει. Εμείς έχουμε την εμπορική συμφωνία θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει την έρευνα και αν αυτοί δεν προτίθενται να ξεκινήσουν μπορούμε εμείς να τους οθήσουμε να ξεκινήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάντοτε εκπλήσωμαι να ακούω όταν υπάρχουν απειλές για κυρώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα εκπλήσωμαι όταν τα αυταρχικά καθεστώτα προστατεύουν τους συνδικαλιστές και τους εργαζομένους. Το βρίσκω πολύ περίεργο διότι οι συνθήκες εργασίες όπως ε, και τα ημερομίσθια δεν πρέπει να καλύπτονται από εμπορικές συμφωνίες αλλά συνδικάτα. Και μας λένε μα δεν υπάρχουν και πολλοί συνδικαλιστές στην Κολομβία οπότε τότε όλοι θα πρέπει να λάβουν το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι όταν βλέπουν με τις διώξεις ε, και τις δολοφονίες όσοι έχουν εναπομείνει πρέπει να πάρουν το βραβείο Ζαχάροφ. Σε μια κατάσταση λοιπόν όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα και πιστεύω ότι ε, εάν μειώναμε τις δολοφονίες κατά 45% θεωρώ ότι δεν επαρκεί αυτό το επιχείρημα διότι όταν είναι η χώρα χώρα όπου διώκονται οι περισσότεροι συνδικαλιστές δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ό,τι κάναμε για τη Σιλάνκα πρέπει να το κάνουμε και για την Κολομβία. Δηλαδή να ερευνήσουμε τι γίνεται στην Κολομβία να διακόψουμε τις συζητήσεις για ελεύθερο εμπόριο διότι ε, βλέπουμε ο, κατόπιν της μελέτης ε, των ε, κοινωνικών επιπτώσεων θα αυξηθεί η βία και θα πρέπει η Ισπανία, και οι Ισπανοί σοσιαλιστές να πάψουν να προασπίζουν τα συμφέροντα των Ισπανικών επιχειρήσεων αντί να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριο κύριος ε, Ζαρβίλ από το ε, κόμμα των Ευρωπαίων ε, Συντηρητικών και πάλι θα μιλήσω τσέχικα. Πρωτού όμως κάνω την ερώτησή μου θα πρέπει να αναφερθώ και να αμφισβητήσω τα στατιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν. Διότι εγώ αν δολοφονόμουν τώρα δεν θα θεωρώμουν σαν ευρωβουλευτής στις στατιστικές αλλά σαν ε, τσέχος και το ίδιο ισχύει για τους συνδικαλιστές. Όταν μιλάμε για θύματα της βίας στην Κολομβία διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί και μπορεί να τριθεί. Οπότε θα ήθελα να ξέρω πόσο έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν πέντε χρόνια ή πριν 10 χρόνια. Αν υπάρχει μία σαφής και αισθητή ε, ε, βελτίωση πιστεύω ότι κάτι τέτοιο ε, ισχύει και θα ήθελα να ξέρω σε τι τιμές βασίζονται, βασίζονται οι κολομβιανοί πολίτες δηλαδή τι θα είχαν, ποια θα ήταν η κατάστασή τους αν δεν είχε υπάρξει αυτή η συμφωνία προτιμήσεως ε, διότι αν πρέπει κανείς να προσπιστεί ορισμένους ε, θα πρέπει εμείς κάτι να κάνουμε διότι συμφωνώ με τη συνάδελφο ότι η κατάσταση αυτή ε, μοιάζει με την περίπτωση της Σρι αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αποσύρουμε την προτίμηση δεν συμφωνώ για το θέμα της Κολομβίας και νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε. Ο Ρίτσαρτ Χάουι τώρα. Καταρχήν, για την Κολομβία θέλω να έχουμε καλές σχέσεις και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα υπογράψουμε μαζί τους μια συμφωνία αλλά τώρα δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή διότι δεν πιστεύω ότι ε, ε, όταν ε, υπάρχουν 60% δολοφονιών και 98% ατιμερησία υπάρχει δικαιοσία. Υπάρχουν συνεχείς απαγωγές και δολοφονίες και αυτό δεν αντικατοπτρίζει χρηστά ανθρώπινα ανθρώπινα ε, Έχουμε 2.600 περιπτώσεις δολοφονιών συνδικαλιστών και περιστατικά και ε, έχουν εντοπιστεί στην, ε, κολονία, στην Κολομβία και μας παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο. Ε, πόσες εξ αυτών των περιπτώσεων έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και έχουν υπάρξει διώξεις σχετικές. Θα έπρεπε εάν υπάρχει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου νομίζω ότι σέβεται κανείς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν βλέπω ποια είναι η διαφορά. Και επίσης ο τελευταίος ομιλητής όταν μιλάμε για 50 σελίδες παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητάμε ε, να γίνει μία εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς δεν συνενέσατε ε, και τα αναφέρει η Βαρόνια Άστον στην επιστολή της και δεν τα δέχεστε ε, θα έπρεπε να έχουμε ε, μία ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε περίπτωση που δεν γίνεται σεβαστή να υπάρχει άρση των, ε, της συμφωνίας διότι διαφορετικά γιατί μας προτείνεται να συνενέσουμε σε μία τέτοια προτιμησιακή συμφωνία η κυρία Λάτφορντ από τους Πρασίνους ε, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο των αρχών και ε, η ε, Κολομβία να σεβαστεί τις αρχές διότι εάν υπάρξει συμφωνία ελευθέρου εμπορίου πιστεύω ότι όχι μόνο θα είναι λάθος να ανταμείψουμε την Κολομβία αλλά θα υπονομεύσουμε και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι ε, δεν έχουμε πιστεί ότι η Κολομβία στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ακούσει για βία, για διωγμούς και έχω ε, μία επιστολή μπροστά μου από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όπου λέγεται ότι υπάρχει στην Κολομβία μεγάλη ανησυχία διότι συνεχίζονται οι δολοφονίες και ε, ε, από το σύνολο περίπου 60 δολοφονιών συνδικαλιστών 48 το 2008 ήταν από την Κολομβία. Θα ήθελα λοιπόν ο, ο πρέσβης να μας πει α, ε, πόσοι ε, υπάρχουν ε, ακόμη εργαζόμενοι οι οποίοι εκπροσωπούνται στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ακούω ότι είναι μόνο 4%. Έχουμε ήδη ζητήσει να υπάρξει μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά αν δεν το επιτύχουμε ε, δεν θα έπρεπε μόνο να ε, αποσύρουμε το προτιμησιακό καθεστώς αλλά και τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Κύριε Πρόεδρε, ε, ε, βρίσκω αξιοπερίεργη την, ε, τη θέση του κυρίου Βαλτεράμα, ο, ο οποίος προσπαθεί να συγκαλύψει τις δολοφονίες των συνδικαλιστών, διότι το ποσοστό λέει των ε, ε, συνδικαλιστών που σκοτώθηκαν ήταν μικρότερο από το σύνολο συνδικαλιστών στην κοινωνία της Κολομβίας. Ενώ συστηματικά υπάρχει διωγμός των ε, εργαζομένων προσπαθούν να οργανώσουν τους συνανθρώπους τους και τους υπολείπους εργαζομένους στην Κολομβία και σκοτώνονται, δολοφονούνται για, διότι προσπαθούν να τους οργανώσουν από ε, μέτρα εκφοβισμού και ε, προσπαθίας να υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των ε, εργαζομένων. Υπάρχει στρατιωτική και παραστρατιωτική εμπλοκή και ο πρέσβης δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα αυτό. Τέλος, ε, δεν αναφερθήκαμε εδώ εις ε, την ε, διεθνική συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι οργανώσεις των της κοινωνίας των πολιτών λέγουν ότι το κράτος συμβάλλει στη βία αυτή και είναι σοβαρές κατηγορίες οι οποίες πρέπει να διαρευνηθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σκηνικό που εμφανίζεται μέσα από αυτή την συζήτηση είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, αλλά κάποια πράγματα μου φαίνονται σαφή. Πρώτον, η Κολομβία εκπροσωπεί ένα είδο ε, μαύρη κοιλίδα μη ειρηνευμένη περιοχή τη Λατινική Αμερική. Τα ποσοστά βία εκεί είναι απαράδεκτα. Δεύτερον, υπάρχουν γκρίζε ζώνε σε ό,τι αφορά τη δράση των αρχών. Όχι τόσο τη επίσημη κυβέρνηση αυτή καθεαυτή, αλλά του συνόλου των αρχών, τοπικών αρχών και περιφερειακών συμπεριλαμβανομένων. Τρίτον, τα δεδομένα είναι αυτά που ακούσαμε. Είναι η πραγματικότητα. Το 60% των συνδικαλιστικών των συνδικαλιστών που θανατώνονται στην, ε, στον πλανήτη μα, ε, δυστυχώ χάνουν τη ζωή του στην Κολομβία κατά κύριο λόγο. Πρέπει λοιπόν το ζήτημα τη Κολομβία να το δούμε ίσω παράλληλα με την υπόθεση τη Σρι Εκεί αντιτίθεμε στην αναστολή του προγράμματο GSP Συν, αλλά θα πρέπει να σταθμίσουμε το κατά πόσο να εμεί δρούμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά για παρόμοιε χώρε. Γιατί στα πλαίσια του προγράμματο GSP Συν ε, έχουμε ξεκινήσει και τις διαπραγματεύσει για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Εδώ λοιπόν πιστεύω, όπω νομίζω και όλε οι υπόλοιπε πολιτικές ομάδες, ότι δεν πρέπει να πάρουμε μια πρωτοβουλία που να ξεπερνά τα πλαίσια της συζήτησή μα. Και ίσως να ζητήσουμε και προφορική εξαίρεση από την πλευρά τη Επιτροπή μα για να έχουμε στη Σύνοδο τη Ολομέλεια του Φεβρουαρίου του Μαρτίου ε, διάλογο για το θέμα αυτό και στην Ολομέλεια. Δηλαδή να δώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο στο ζήτημα και να αναβαθμίσουμε θεσμικώ την εξέταση τη Κολομβία. Να εμβαθύνουμε και να αναλάβουμε και τι ευθύνε που μα αρμόζουν. Ε, και ε, επίσης να δεσμεύσουμε και τον νέο επίτροπο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα. Και εδώ θα πρέπει πραγματικά να έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ένα ερώτημα και μετά να δούμε τι συμπεράσματα θα προκύψουν. Ευχαριστούμε, το καταγράφουμε αυτό που είπατε. Δεν είναι καθόλου κακό να έχουμε προφορική ερώτηση για το θέμα αυτό. Τέλο, ο κύριο Μενέντε. σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έλεγα στον κύριο Μάρτιν ότι δεν έχει καταγραφεί η ε, δική του έτσι να πάρει το λόγο. Υπάρχει αντικειμενικά ένα σύνολο δεδομένων που αποδεικνύουν ότι έχει γίνει καταστρατήγηση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία. Και υπάρχουν δύο απόψεις. Αυτοί που πιστεύουν ότι συνεχίζει να γίνεται καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την άμεση ή έμεση ε, συνεργασία, συνωμοσία της κυβέρνησης, κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη, αλλά άρχισε να ενεργεί σιγά σιγά η κυβέρνηση για να μπορέσει να σταματήσει αυτή η καταστροφική κατάσταση του παρελθόντος. Εγώ είμαι υπέρ του της Δευτέρας, ε, μεταξύ των αυτών που σκέφτονται ότι ισχύει η δεύτερη, δεύτερη άποψη. Πιστεύω ότι η νέα στάση της κυβέρνησης της Κολομβίας προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση και πιστεύω ότι θα μπορούσε να συναυθεί αυτή η σύμβαση με συστήματα εποπτείας για να είμαστε ε, να, για να συμπεριλάβουμε τους πάντες αντί να αποκλείσουμε τους πάντες. Πιστεύω ότι έχει αποδείξει η κυβέρνηση της ε, ε, Κολομβίας ότι μπορεί να κάτι για να βελτιωθεί το μέλλον. Δεν λέω τίποτα άλλο γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά πιστεύω ότι είπα τα πάντα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν πήρα υπόψη μου τη ζητήση το λόγο, κύριε Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο πολύ γρήγορα ερωτήματα, επειδή περνάει ο χρόνος. Ο τελευταίος από τους επισκέπτες μας, από την Ένωση Δημηχάνων και Επιχειρηματιών, μας απαρίθμησε έναν εντυπωσιακό κατάλογο με τις προσδοκίες του για να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος και να προστατευτούν οι πρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Να ρωτήσω, γιατί αυτά είναι απλές προσδοκίες, γιατί δεν υλοποιούνται όλα αυτά. Μήπως δεν υπάρχει κυβερνητική στήριξη, τι τους εμποδίζει να επιδιώξουν τους στόχους αυτούς. Και το δεύτερο ερώτημά μου απευθύνεται στον ε, πρέσβη. Και αφορμή λαμβάνω και από τα όσα είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Εάν πράγματι έχει βελτιωθεί αξιοσημείωτα η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, γιατί η κολομβιακή κυβέρνηση δεν ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια εντελεχή και διεξοδική έρευνα τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία, ώστε να έχουμε μια μερόληπτη τοποθέτηση για το τι συμβαίνει με το θέμα αυτό και να έχουμε και ξεκάθαρου όρου περιγραφή τη κατάσταση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ναι, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και την Επιτροπή όμως, πριν δώσω τον λόγο στους προσκεκλισμένους μας και ο χρόνος μας εξαντλείται. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω στην Επιτροπή περισσότερα από τρία λεπτά. Αλλά υπάρχουν ζητήματα στα οποία ήθελα ίσως να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προϋποθέσεις για το πρόγραμμα GSP συν γίνονται σεβαστέ από την Κολομβία. Γιατί να μην υπάρξει έναρξη μια νέα φάση. και αυτό το έθεσαν τουλάχιστον δύο από τα μέλη της Επιτροπής μας. Το λόγο έχει λοιπόν ο κύριο Ζωά Γκέρ Μαχάδου, Γενικός Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ που είστε μαζί μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω εκτός μικροφώνου. Πρέπει να πω για την όλη κατάσταση ότι οι ανταλλαγές και η συζήτηση που είχαμε σήμερα το απόγευμα έχουν ε, ήδη εξεταστεί σε επίπεδο πληροφόρηση από την Επιτροπή. Έχουμε λάβει στοιχεία από διαφορετικέ πηγέ για το πώ η Κολομβία υλοποιεί το πρόγραμμα GSPC και κυρίως σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει της ε, που απορρέουν από τι ε, ανάλογε συμβάσει. Η, καθο... η βασική γραμμή που ακολουθήσαμε σε όλες μας τις εκτιμήσεις, αποτιμήσεις και εξολογήσεις βασίστηκαν στα στοιχεία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών φορέων. Η κατάσταση στην Κολομβία σαφώ δεν είναι ιδανική. Πολλά θέματα προκαλούν ανησυχίες, αλλά επίσης είναι βέβαιο ότι έχει επιτελεστεί πρόοδο από την κυβέρνηση για την υλοποίηση και την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντόπισαν κάποιοι από τους φορείς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κολομβιανή κυβέρνηση έχει περάσει εντατικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, αναζη... και είναι η άποψη της Επιτροπής ότι ο διάλογος αυτός οθεί την ε, Κολομβιανή κυβέρνηση να ακολουθήσει μια πιο δραστήρια στάση, ενεργή συμμετοχή και να περάσει σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά προβλέπονται και από το καθεστώ του προγράμματος GFPC. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση της κατάστασης. Η κατάσταση τώρα της Σρι Λάγκα είναι ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Εκεί δεν υπήρξε καμία συνεργασία, καμία συζήτηση με την Επιτροπή, είτε πριν είτε κατά της, ε, ε, τη διαδικασία ερεύνης που ξεκίνησε και θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο περιπτώσεις μεταξύ τους. Διότι είναι πολύ διαφορετικά τα πολιτικά σκηνικά στην μια και στην άλλη. Οι κατηγορίες για βία είναι πολύ διαφορετικές στη μια περίπτωση και στην άλλη. Έτσι λοιπόν η πολιτική μας βλέπουμε να δίνει αποτελέσματα, συγκεκριμένα αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι η Κολομβία θα πρέπει να έχει άλλη μια ευκαιρία να μπορέσει να ε, προσπαθήσει να επιδιώξει τους στόχους των συστάσεων του ILO και της, του ΟΗΕ, e, όπως απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτή την πολύ συγκεκριμένη απάντηση στις ερωτήσεις και τα σχόλια που απευθύνθηκαν προς εσάς, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα φτάνουμε προς την λήξη της συζήτησής μας να δώσω το λόγο στους βασικούς μας προσκεκλημένους, στην ίδια σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν αρχικά. Ξεκινάμε από τον κύριο Φράνκο. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω το εξής το ανακοινωθέν στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Βάνεγκας όπου λέει ότι σε δεν μου επιτρέπει να λάβω το λόγο εξ ονόματός του είναι ανακοινωθέν της 4ης Μαΐου του προηγούμενου χρόνου όταν είχαμε έρθει εμείς εδώ. Προφανώς από τότε που άρχισε την παρέμβασή μου είπα ότι δεν εκπροσωπούμε καμία συνομοσπονδία. Είπα όμως ότι άλλαξε τη στάση της συνομοσπονδίας συνδικάτα μας σε σχέση με την συνθήκη στο τέλος του 2009. Άρα, καλό είναι να το διευκρινίσουμε αυτό. Διότι βλέπω ότι σήμερα κάποιος κατέβασε το ανακοινοφέν αυτό από το ίντερνετ και το έφερε εδώ, αλλά του άλλαξε η ημερομηνία. Όταν πρόκειται για να πει κάποιος κάτι αντιφατικό στη χώρα μας και κυρίως εκ μέρους της ΚΟΥΤ, αυτό το οποίο κάνει όταν δεν έχει επιχειρήματα είναι να παρουσιάσει εσφαλμένα στοιχεία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε πλειοψηφία ε, στον ιδιωτικό τομέα, στην ΣΕΖΕΤΕ. Ο τομέας τον οποίο εκπροσωπώ είναι πλειοψηφία του συνδικάτου. Και οτιδήποτε γίνει σε σχέση με εμπορικές ε, συμφωνίες, θετικό ή αρνητικό, αφορά 14 εκατομμύρια εργαζόμενου, 96 από τους οποίους δεν είναι μέλη συνδικάτων. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι στην περιοχή στην οποία ζω εγώ εδώ και 25 χρόνια με... και είμαι μέλος της συνδικαλιστικής οργάνωσης των παραγωγών ε, μπανάνας έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις αλλά υποφέραμε από την ε, ε, βία το δεκαετίας του 90 που προκάλεσαν οι επαναστάτες του LRVM. Κανένας όμως μέχρι σήμερα συνδικαλιστής τα τελευταίο χρόνο δεν έχει συλληφθεί αφαίρετα ή δεν έχει δολοφονηθεί. Πρέπει να πω ότι κάναμε απεργία και έγινε σεβαστή από τους εργαζομένους. Έχουμε συζητήσει με τους εργοδότες και αναγνωρίστηκε και από τους συναδέλφους που είναι μέλη της ΚΟΥΤ και από τους εργοδότες η στάση μας. Επίσης θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο σας έχει διανεμηθεί όπου ορίζομαι εκπρόσωπος εγώ. Πράγμα το οποίο είναι χαστούκι προς αυτούς οι οποίοι είπαν ότι εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος. Έχει υπογραφεί από έναν συνάδελφο, ο οποίος σήμερα είναι υποψήφιος για τις βουλευτικές εκλογές. Αυτό που αναφέρεται στο εγγραφό είναι μία απεργία η οποία οργανώθηκε και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν αντίθετοι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στο έγγραφο αυτό. Αυτή είναι μία ευκαιριακή, ε, ένας ευκαιριακός τρόπος αντίδρασης των συντρόφων της ΚΟΥΤ. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι με τη στάση μας να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα. Είμαστε ε, επειδή μας πονάει αυτό το οποίο γίνεται στη χώρα μας και μας πονάει το ότι υπάρχουν τόσ θύματα ανοιχτή σε οποιαδήποτε συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Βανταγκάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι Τα τρία συνδικάτα ε, ενωμένα στα πλαίσια της νομοσπονδίας ζητήσαμε από την διεθνή κοινότητα και βάσει των διαφόρων αναφορών που υπάρχουν από διεθνείς οργανώσεις και από την Amnesty International και από αυτούς οι οποίοι τώρα τελευταία έκαναν μία έκθεση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει να πω ότι δόθηκαν και κονδύλια κοινοτικά και δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο οι συνδικαλιστές αλλά οι φοιτητές, οι δικαστές, δημοσιογράφοι, Όλοι πρέπει να πω ότι σήμερα υφίστανται πιστέψεις. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μία διεθνής εκστρατεία υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των Κολομβιανών. Θέλουμε μία τέτοιου είδους συμφωνία να μην υπογραφεί με την κυβέρνηση της Κολομβίας. Έχω την εντύπωση ότι ο πρέσβης Κύριε Στροχίγιο, είπα ότι είναι διατεθειμένος να δεχθεί όλους όσους θέλουν να κάνουν επισκέψεις ή να δεχθεί οποιαδήποτε έρευνα για οποιαδήποτε θέμα. Γιατί δεν μίλησε για αυτή την δική μας την ε, ε, σύμβαση, την ΣΕΧΕΤΕ πλούς. Θα ήθελα να εκφράσει τη βούλησή του και η κυβέρνηση να γίνει πριν να υπογραφεί το τέλε μία εκ των προτέρων μελέτη. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι στην περίπτωση ότι μάλλον στην Κολομβία όταν οι εργαζόμενοι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κατάσταση σκλαβιάς για κάποιους και ξέρετε τι συνέβη με την περίπτωση κάποιων εργαζομένων που δούλευαν στο ζαχαροκάλαμο που έπρεπε να εργαστούν για κάποιες επιχειρήσεις χωρίς να έχουν καμία ε, σύμβαση και έχουμε περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι εργάζονται ε, βάσει κάποιων συμφερόντων και χωρίς αμοιβή ή την χάνουν θύματα εγκα... εκμετάλλευσης από κάποιους συνεταιρισμού, διότι τους δίδεται ένα μικρό καταποκοπήν ποσό για να καταβάλουν αυτοί όλα τα, για να πληρώσουν αυτοί τελικά όλες τις δαπάνες που κάνουν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταγγείλουμε. Πρέπει να πω ότι έκαναν αυτοί οι ίδιοι απεργία διότι βαρέθηκαν να δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες και πρέπει να πω ότι για να μπορέσουν να, για να προστατεύσουν τη ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους χρειάστηκε να επέμβουν ξένες δυνάμεις. Υπάρχει λοιπόν μία κουλτούρα κατά των συνδικάτων ε, στην ε, Κολομβία. Να απαντήσω για την ε, ατιμορρησία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελία, η ατιμορρησία φτάνει σε ποσοστά 98% και με αυτός τους ρυθμούς θα πρέπει να περιμένουμε δεν ξέρω πόσα χρόνια για να δούμε από τις 2.000 2.700 επιστάσεις που εκκρεμούν ε, θα ε, δικαιωθούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ επικοδομητική, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα πλέον έχουμε γνώση του πώς έχει κατάσταση στην Κολομβία. Και θα πρέπει να εξετάσουμε και τις δικές μας τις θέσεις ως προς τις παραχωρήσεις ή όχι του δικαιούχου χώρας του προγράμματος GPS SIN για την Κολομβία. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, προσκεκλημένους μας και κυρίως τους βασικούς ομιλητές. Εδώ κλείνει η συζήτηση για σήμερα. Ε, Προχωρούμε τώρα στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Σας παρακαλώ να ησυχάσετε. Και όσοι θέλετε να φύγετε από την αίθουσα, κάντε το σιωπηρά. And please avoid speaking. Παρακαλώ αποφύγετε τις ομιλίες κάτω στην αίθουσα. Please. Please, those who are Παρακαλώ, όσοι βγαίνετε από την αίθουσα, φροντίστε να το κάνετε αυτό λίγο πιο γρήγορα. Φτάνουμε προς το τέλος της συνεδρίασής μας, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ. Πηγαίνουμε τώρα στο σημείο 12, νέες εξελίξεις στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Το θέμα αυτό είναι από την ευθύνη της Επιτροπής ΙΜΚΟ Τώρα εξετάζουμε ένα σχέδιο έκθεσης για το γνωμοδότηση για, την... για το θέμα της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Εδώ η συντάκτη της γνωμοδότησης είναι η Μαλγκορθάτα Χάντλικ για το ΕΛΚ. Να θυμίσω ότι το μέσο των δημόσιων συμβάσεων έχει γίνει ένα σημαντικό σκέλος ε, των εμπορικών πολιτικών, αν και ο τομέας αυτός δεν περνά στο πολυμερέ σύστημα, δεν εμπίπτει στο πολυμερέ σύστημα του ΠΟΕ. Απλώ ορίζεται από τι κυβερνητικέ συμφωνίε για τι δημόσιε συμφωνίε, την GPA, η οποία είναι ούτω ή άλλω πολυμερή από τη φύση τη. Οι εμπορικά σημαντικέ χώρε, όπω η Κίνα, δεν συμμετέχουν όλε στο GPA. Ενώ είναι αναμενόμενο από καιρό η αναθεώρηση του συστήματο αυτού αλλά για την ώρα φαίνεται να έχει παγώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση για το θέμα από πέρσι τον Οκτώβριο. Σε αυτό το πλαίσιο καλό είναι να θυμόμαστε ότι η εσωτερική αγορά και οι εμπορικές της σχέσεις είναι βεβαίως άρρηκτα συνδεδεμένες. Εμείς, ως Επιτροπή Υπεύθυνη για τα θέματα διεθνούς εμπορίου, Παρακολουθούμε τι παρέμβαση έχουν γίνει στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων ως τώρα. Πώς χειρίζονται το θέμα αυτό οι εσωτερικές αγορές και βεβαίως αναγνωρίζουμε την επίδρασή τους και στο δικό μας τομέα. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση αυτή και θα δώσω το λόγο κατευθείαν στην εισηγητριά μας. Ε, Ευχαριστώ. Με τα μεγάλη χαρά ε, ε, λαμβάνω το λόγο σχετικά με το θέμα αυτό και πρέπει να πω ότι ε, είχε γίνει προηγουμένως μία ακρόαση σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και ήθελα να δω τι γινόταν ε, και εάν χρειάζονται ε, άλλες νέες ε, άδειες. Πρόκειται για θέμα εσωτερικής αγοράς και γι' αυτό ο εισηγητής θα ασχοληθεί με αυτή την πτυχή. Μέχρι στιγμής είχαμε ασχοληθεί με εθνικά θέματα και γι' αυτό αυτό πήγα σε αυτή την ακρόαση και θα μπορούσα να σας πω ποια θέματα έθιξα. Η αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ανοιχτή και κάθε χώρα μπορεί να συμμετέχει εις τους δημόσιους διαγωνισμούς και εις τις εθνικές συμφωνίες. Η αγορά των δημοσίων συμβάσεων τις τρεις χώρες δεν είναι πάντοτε ανοιχτέ στον ίδιο βαθμό στις ευρωπαϊκές εταιρείες και ενώ έχουμε συμφωνίες με ε, εμπορικούς εταίρους αυτή η αμοιβαιότης δεν είναι εγγυημένη και πολλές ε, επιχειρήσεις στην Ευρώπη μιλούν για ε, δυσκολία προσβάσεως σε αγορές τρίτων χωρών. Όντως η κατάσταση ε, είναι δύσκολη ε, σχετικά με τις ε, τρίτες χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες δημοσίων συμβάσεων διότι μας περιορίζουν ακόμη περισσότερο όσον αφορά την πρόσβαση στην εσωτερική τους αγορά. Παραδείγματος χάρη, η Κίνα τελευταίως έχει εισάγει ένα σήμα διαπιστεύσεως για τα νέα καινοτόμα προγράμματα προγράμματα και ε, ευνοεί τα ε, διαπιστευμένα προϊόντα ε, για τις δημόσιες συμβάσεις της. Και αυτό βέβαια έχει σχέση με τοπικές κινέζικες εταιρείες, οπότε φοβόμαστε ότι μέσω της καταγραφής και της διαπιστεύσεως μειώνονται οι δυνατότητες μας και θα πρέπει να εστιαστούμε ε, σε πολυμερείς συμφωνίες όπως παραδείγματος χάρη τον ΠΟΕ όπου υπάρχουν διαπραγματεύσεις σχετικά με το θέμα αυτό αλλά είναι δύσκολες ε, και μακρόπνος και θα πρέπει να περιμένουμε να τελεσφορήσουν. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει αυτές τις διαπραγματεύσεις χωρίς να ξεχνά τις φιλοδοξίες μας. Βέβαια, το άνοιγμα αυτών των αγορών θα πρέπει να ενθαρρύνει και τους ομολόγους μας να ανοίξουν τις δικές τους αγορές. Δηλαδή, όσες ε, χώρες ε, δεν ωφελούνται από την αμοιβαιότητα και δεν υπάρχει ανοιγμά θα μπορούν ε, στο μέλλον εφόσον είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να επιτρέψουν περιορισμούς διότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εταιρείες να, ε, να ανταγωνίζονται μαζί μας χωρίς εμείς να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τις εταιρείες τους στις δικές τους αγορές. Άρα η ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να ε, υποδηλώσει ότι ε, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι εντός παρενθέσεως dumping και προστατευσισμού στις δικές μας αγορές. Ε, είναι κάτι επί του οποίου θέλω να ερευνήσω το θέμα περαιτέρω και θα πρέπει να το θυμόμαστε. Θα ε, περιμένω τα σχόλιά σας και σας υπενθυμίζω ότι η ε, προθεσμία για τροπολογίες είναι 29 Ιανουαρίου μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Νομίζω ότι τώρα θα έχουν τον λόγο οι εισηγητές και ξεκινάει ο κύριος Γιώργη Κούτας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν σημαντικές, ε, σημαντικά στοιχεία που θα έπρεπε να περιληφθούν στην έκθεσή της. Δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχουν αρχές πρασίνων δημοσίων συμβάσεων και δυνατότητος να χρησιμοποιηθούν οι δημόσιες συμβάσεις για να προωθηθεί η αηφόρος ανάπτυξη και επειδή σήμερα έγινε μια μακριά συζήτηση νομίζω ότι είναι πολύ βασικό να περιληφθεί στο σχέδιο της γνωμοδότησης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των κοινωνικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως καταγράφονται εις την διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε το μηχανισμό κατά της διαφθοράς. Στον τομέα των διεθνών συμβάσεων στα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες για επίτευξη διαφθοράς και για περιστολή των δημοσίων δαπανών. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος σκιώδης ο οποίος θέλει να αναφερθεί στο θέμα αυτό. Τότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Έρικ Νότεμπαου από την Γενική Διεύθυνση ε, Αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε με αυτά τα οποία είπε η συγκήτρια διότι ε, όντως οι διεθνείς ε, διαπραγματεύσεις για τις δημόσιες συμβάσεις είναι δύσκολο θέμα ιδίως διότι πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια ανοιχτή αγορά που δεχόταν όλες τις ε, ε, προσχωρήσεις ε, ενδιαφερομένων. Και όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, οι χώρες αυτές δεν είναι εξίσου ανεχτές και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διατυπώσει πρόταση για να υπάρξει μία πιο αυστηρή εφαρμογή της αρχής της ε, αμοιβαιότητος, δηλαδή στην πρόταση που είχαμε υποβάλει το Φεβρουάριο 2009 αναφερθήκαμε ε, σε περιορισμούς για τις αμερικανικές εταιρείες από τις είπα δηλαδή ή στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων διότι εις ε, την Αμερική υπάρχει μία αρχή set aside for, ε, ε, για αμερικανικές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αποκλειστική χρήση και άρα δεν ισχύει το ίδιο στην Ευρώπη. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι στην τωρινή οικονομική κρίση διεθνώς υπάρχουν ε, περιορισμοί κατά τρόπον ώστε τα, οι δημόσιοι πόροι να καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες των εθνικών επιχειρήσεων αλλά πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επιμείνουμε στην αρχή ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοιχτή οικονομία αλλά όταν αντιμετωπίζουμε αντίθετες μεθόδους δεν θα διστάσουμε και εμεί να χρησιμοποιήσουμε περιοριστικές μεθόδους. Ε, όπως σας είπα συμφωνώ απολύτως με την εισηγήτρια την κυρία Χάντλικ και ε, με τα σχόλιά της. Κάποιος άλλος ζητά το λόγο πριν δώσω το λόγο στην κυρία Χάντλικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια για το σχέδιο γνωμοδότηση. Νομίζω υπάρχει μια γενική παρατήρηση, όπω είπε και ο σκιώδη εισηγητή, και θα εξετάσουμε με σοβαρότητα τι τοπολογίε του. Πρέπει να έχουμε ίσως λίγο πιο καταμένη συζήτηση στην επόμενη συνεδρίασή μα. Σας ευχαριστώ πάντω πάρα πολύ. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. referred to and also the votes in this Θα ψηφίσουμε σε αυτή την Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 15. Να σας ενημερώσω επίσης ότι τα πρακτικά από τις συνεδρίες των συντονιστών την πρωινή ήδη έχουν διατεθεί, μοιράζονται στο βάθος της αίθουσας και βάσει της τακτικής μας διαδικασίας θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εφόσον δεν υποβληθούν ε, αντιρρήσεις ή σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο 15. Ενδιάμεση επανεξέταση των εγγράφων γεωγραφικής και θεματικής στρατηγική δύναμη του κανονισμού 1905 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εδώ έχουμε ανταλλαγή απόψεων για την ομοδότηση με αρμόδια επιτροπή, την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Δικός μας συγγετή είναι ο κύριος Μάρτιν από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Γιατί η Επιτροπή Ανάπτυξη αποφάσισε να συντάξει έκθεση ιδέε πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Και η δική μα ε, Επιτροπή αποφάσισε με τη σειρά τη να σχολιάσει γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να χρηματοδοτήσει χώρες βάσει του κανονισμού του μηχανισμού μάλλον χρηματοδότησης, αναπτυξιακής συνεργασίας Βάσει των εγγράφων που προαναφέραμε, είναι τα βασικά εργαλεία του μηχανισμού αυτά γιατί αποτελούν πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών πολιτικών, των πολιτικών συνεργασίας. Υπάρχουν εργαλεία για την διαχείριση, την αναθεώρηση και την αποτίμηση των ε, ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κύριε Μάρτιν, έχετε το λόγο για αυτήν την ομοδότηση. Ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά έχω πολύ λίγα να πω. Θα, θα αφήσω λοιπόν ε, την εξέλιξη της συζήτηση στα χέρια και στη σοφία των μελών της Επιτροπής. Όπως είπατε τα έγγραφα αυτά γεωγραφικής και θεματικής στρατηγικής είναι καθοριστική σημασία για το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα πρέπει να παρουσιάζουν συνοχή με άλλα μέσα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή συζητήσαμε και το πρωί ότι το εμπόριο μπορεί να είναι μια κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη του εμπορίου και την οικονομική αύξηση, πρέπει το εμπόριο να το βλέπουμε ως, μέρο ενός, μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου, για την αναπτυξιακή συνεργασία. Και προκειμένου να διευκολύνουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν εμπορικές συναλλαγές. Οι φτωχότερες χώρες του κόσμου χρειάζονται περισσότερη πρόσβαση στις δυσυνοριακές αγορές. Και για να μπουν σε αυτές τις αγορές πρέπει να έχει συμφωνηθεί προηγουμένω στρατηγική, όπω αυτή του Hong Kong το 2007 ή το πρόγραμμα Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο. Η μόνη πτυχή του DCI που πρέπει εδώ να προσθέσουμε είναι η διάσταση του Aid for Trade. Και μέσω της έκθεσης της Επιτροπής ΔΕΒΕ θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, λεπτομερείς πληροφορίες για το πώ η ανάλογη δημοσιονομική γραμμή δαπανάται και τι γίνεται με τις υπόλοιπες πολιτικές που υλοποιούμε βάσει του οργάνου DCI. Για την ώρα αυτά έχω να πω κύριε Πρόεδρε για το θέμα αυτό και επαναλαμβάνω το ζήτημα που το θέτω στην κρίση των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής. Πρόεδρος, η Επιτροπή Ποιο παίρνει το λόγο εκ μέρου τη Επιτροπής. Κύριε Σίμεκ, κύριε Λουγκερό, κύριε Πρόεδρε, λέγομαι Ροτ ε, από τη Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ, όπου εργάζομαι, και είμαι συντονιστή τη ε, διαδικασία ενδιάμεση επανεξέταση εκ μέρου τη Γενική μα Διεύθυνση. Αληθεύει ότι υπάρχουν εδώ στοιχεία εμπορικά στα έγγραφα του DCI και στα στρατηγικά έγγραφα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απαντήσουμε στα σχόλια που είχε κάνει το Κοινοβούλιο μετά την προηγούμενη περίοδο του προγραμματισμού μας και προκειμένου να συνδυάσουμε οριζόντια ζητήματα και να γίνουν οι μικρές μας δημοσιονομικές γραμμές πιο αποτελεσματικέ. Το Aid for Trade έχει πολύ μικρή δημοσιονομική γραμμή, αλλά προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τι πτυχέ του Aid for Trade στο ευρύτερο πλαίσιο των πακέτων. Το άλλο στοιχείο που επεξεργαζόμαστε και που κανείς δεν έχει αναφέρει ακόμη είναι το εργαλείο για τις βιομηχανοποιημένες χώρες. θα πρέπει να δούμε και τη μη αναπτυξιακή μας ε, συνεργασία στο μέλλον, δηλαδή από το 2011 στο 2013. Πάντως αναγνωρίζουμε ότι το εμπόριο είναι κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το σχετικό πρόγραμμα, το Aid for Trade, για να ακολουθήσουμε την πεπατημένη της αναπτυξιακής συνεργασίας. Εάν θέλετε, θα απευθυνθώ στις υπηρεσίες της RELEX και θα τους ζητήσω να σας ετοιμάσουν ένα ενημερωτικό σημείωμα για το πώς ο προπολογισμό του Aid for Trade και το σχετικό πρόγραμμα εξελίσσονται. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ευπρόσδεκτη πρόταση. Θέλει κάποιο το λόγο. Κύριε Μάρτιν, άλλες παρατηρήσεις. Όχι. Θα συμφωνήσω με την Επιτροπή ότι και εμεί ένα τέτοιο ενημερωτικό σημείωμα με χαρά θα το δεχτούμε. Εκτός μικροφώνου πρόεδρος πάλι. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και την έγκριση στη συνάντηση του Μαρτίου. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι η λήξη της συνεδρίασης. Είχαμε μια μακροσκελέστατη συνεδρίαση και συζήτηση. Επόμενη συνεδρίαση στις 8 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο, πριν την επίσημη στις 23 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Στο Στρασβούργο 9 το πρωί. Μην το ξεχάσετε. Θα ξεχάσετε το δείπνο, κύριε, τη βραδιά και θα